Θα ήθελα να σας κάνω πρόταση. Να μας κάνει μια σύντομη εισαγωγή η κυρία Κοπά, παρακαλώ, στην έκθεσή της. Και μετά να ακούσουμε το Γενικό Διευθυντή της ε, Γενικής ε, Διεύθυνσης συγγνώμη, για τη Διεύρυνση να μας παρουσιάσει τη θέση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά δήλωσε πρόθυμος να μας πει και για την έκθεση που ενέκρινε σήμερα για την παρακολούθηση της Κροατίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω θα είχε νόημα να μας μιλήσει αμέσως μετά την κυρία Κοπά, ο Γενικός Διευθυντής. Και μετά να κάνουμε μια κοινή συζήτηση, αν συμφωνείτε. Συμφωνείτε? Καλώς. Η κυρία Κοπά έχει το λόγο, παρακαλώ. Thank you, Mr. My report originates from υπάρχει ανάγκη να σκεφτούμε την διεύνηση ε, μετά τη συνοκορυφή της Κοπενχάγης, να διδαχθούμε από τις παρελθούσες εμπειρίες, να καταλάβουμε καλύτερα που βρισκόμαστε σήμερα και να κάνουμε κάποιες συστάσεις συγγνώμη, για το μέλλον. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να γίνει τώρα ε, σε μια εποχή δινής οικονομικής κατάστασης και ε, κούραση για τις αλλεπάλληλες διευρύνσεις. Εγώ θέλω να τη δω από απόσταση και από μια σκοπιά στρατηγικής ε, τη διεύρυνση, να δούμε ε, ποιες είναι οι διαδικασίες, να τις αξιολογήσουμε και να δούμε ποια είναι η πολιτική συνολικά. Ε, πρόσεξα λοιπόν να μην αναφέρω συγκεκριμένες χώρες, ούτως ώστε να μην χάσουμε την εστίαση από την ίδια την πολιτική και θα συμφωνείτε πιστεύω ότι δεν έχει νόημα να μιλήσουμε για συγκεκριμένες χώρες, γιατί έχουμε συγκεκριμένες αιτήσει εκθέσεις αναχώρα. 20 ε, χρόνια μετά από τη συνοκορυφή της Κοπενχάγης ε, έχουμε μια καλή ευκαιρία και μια και είναι και η Δανέζικη Προεδρία, είναι καλή ευκαιρία να σκεφτούμε τα κριτήρια της Κοπενχάγης, να δούμε πόσο αποτελεσματικά είναι χάρη στην ευελιξία τους, όπως μας σε πρόσφατα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η προϋπόθεση για τις υποψήφιες χώρες να έχουν σταθερούς θεσμούς, ε, εξασφαλισμένη δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα, κράτος δικαίου, ε, λειτουργούσα η οικονομία της αγοράς και να μπορέσουν να αναλάβουν τις υποχρεώσεις της ε, ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο τέλος της διαδικασίας, θα πρέπει να παραμείνει ως προϋπόθεση της ε, πολιτικής διεύρυνσης. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όλοι είναι τέλεια. Στην έκθεσή μου, Φερρυπίν, τονίζω όχι μόνο την ανάγκη να προσαρμόσουμε τα οικονομικά υποκριτήρια ε, με βάση τις πρόσφατες εξελίξεις ε, στον τομέα της οικονομικής διακυβέρνησης, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τις κοινωνικές επιπτώσεις για τις υποψήφιες χώρες και δυνητικές υποψήφιες χώρες. Αυτές οι χώρες θα πρέπει να είναι ικανές να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό και να σέβονται ε, τον κανόνα της δημοσιονομικής σταθερότητας. Επιπρόσθετες προσπάθειες λοιπόν χρειάζονται για μια ε, ομαλή οικονομική ένταξη, για την κοινωνικο-οικονομική σύγκληση, ούτως ώστε να μην έχουν ε, υπερβολικές απώλειες θέσεις ε, απασχόλησης κατά τη διάρκεια αυτής της προσαρμογής. Μην ξεχνάμε παράλληλα ότι το τμήμα τη ελκυστικότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλεται στην, στο μοναδικό συνδυασμό οικονομία τη αγορά με βασικά ε, κοινωνικά κριτήρια, πρότυπα που ισχύουν σε όλα τα κράτη-μέλη. Στην παράγραφο 3, αυτή η κοινωνική διάσταση ε, την έχουμε παραμελήσει στην διαδικασία διεύρυνση. Ε, τα βασικά κοινωνικά πρότυπα είναι σημαντικά, δεν πρέπει να κάνουμε κοινωνικό dumping. Η Κομισιόν θα πρέπει να δει πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το κοινωνικό ντάμπινγκ που γίνεται στις ε, υποψήφιες χώρες. Η έκθεση είναι καλή ευκαιρία για να αντιμετωπίσουμε το βασικό σημείο της αξιοπιστίας της διαδικασίας διαέμπρινσης. Ε, βασικό θέμα που συνδέεται με την αιρεσιμότητα και την αποτελεσματικότητα της σας και την ικανότητα απορρόφησης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρώτο μου σημείο είναι ότι η ευελιξία των κριτήρων της Κοπενχάγης και η νέα ε, τιμοπαράδοτη προσέγγιση της Κομισιόν θα πρέπει να ε, οδηγήσουν σε δύο μέτρα και σταθμά και αδικίες για τις χώρες αυτές. Κάθε χώρα θα πρέπει να κριθεί με βάση τις ικανότητές της και θα πρέπει να πληρεί τα ίδια κριτήρια. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν επιπλέον κριτήρια ε, σε μια συνεχιζόμενη διαδικασία και δεν θα πρέπει να έχουμε υπερβολικές απαιτήσει ε, απέναντι στις χώρες αυτές. Και το λέω αυτό γιατί και στο Κοινοβούλιο ε, από καιρού καιρών βλέπουμε τροπολογίε που ζητάνε από ψήφιε χώρες ε, πράγματα που εμεί οι ίδιοι τα σημερινά μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε και δεν μπορούμε να εκπληρώσουμε. Επομένω, η πραγματική ευθυγράμμιση με το κεκτημένο και τα πρότυπα τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι η βασική αρχή που μα καθοδηγεί, χωρί να ε, ξεχνούμε βεβαίω τι ιδιαιτερότητε τη κάθε χώρα. Ε, θα πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Είναι ο πρώτος τρόπος για να είμαστε αξιόπιστοι. Ε, άλλος τρόπος είναι για να έχουμε, και, ε, να έχουμε διαφάνεια και προβλεψιμότητα στην όλη διαδικασία. Είμαι υπέρ της δια, ε, πρόθεσης της Κομισιόν να την κάνει... να την α, συνδυάσει με κάποια κριτήρια ορόσημα. Ε, και σε κάθε φάση της διεύρυνσης θα πρέπει να πληρούνται αυτά τα benchmark, αυτά τα ορόσημα, αυτά τα κριτήρια. Θα πρέπει να είναι δίκαια και να τα προσμετρούμε αντικειμενικά θα πρέπει οι χώρες υποψήφιες να ξέρουν τις προϋποθέσεις ε, στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων και θα πρέπει να ξέρουν τι πρέπει να κάνουν ούτως ώστε να γίνουν οι δυνητικά υποψήφιες χώρες, τι πρέπει να κάνουν και να γίνουν υποψήφιες χώρες. Ακριβώς γι' αυτό θέλω ε, οι εκθέσεις προόδου να είναι πιο ε, προβλέψιμες, ούτως ώστε να χρησιμοποιηθούν ως χάρτης πορεία ω οδικό χάρτη για τι υποψήφιε χώρε. Χαίρομαι για τη νέα μέθοδο τη Κομισιόν που δίνει προτεραιότητα θέμα, ε, σε ζητήματα όπω ε, θεμελιώδη δικαιώματα, ε, δικαιοσύνη, εσωτερικέ υποθέσει, καθώ και ελευθεροτυπία. μέσω της νομοθεσίας και στην πράξη. Η αυστηρή ερωσιμότητα όμω δεν μπορεί να οδηγήσει πουθενά αν δεν υπάρχει αξιοπιστία τη υπόσχεση τη ένταξη. Γι' αυτό είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο να επαναδιατυπώσει την δέσμευση και να κρατήσει τις υποσχέσεις που έκανε ότι θα ενταχθεί κάποιος όταν πληρεί τα κριτήρια, αλλά και να μην δίνει υποσχέσεις όταν δεν μπορεί να τις κρατήσει. Να τις κρατήσει. Θα πρέπει η χώρα λοιπόν να ξέρει εκ των προτέρων που βαδίζει. Και τη στιγμή που ετοιμάζεται η γνωμοδότηση για μια χώρα, θα πρέπει να ξέρουμε τι μέλη γενέστε. Αυτό δεν σημαίνει ότι μετά θα πρέπει να ξεχνάμε την, ε, τις ιδιαιτερότητες της ε, χώρας. Θα πρέπει τη στιγμή που συμφωνούμε για την έναρξη των διαπραγματεύσεων ε, να δούμε τι προσαρμογές πρέπει να κάνουμε και η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτως ώστε να μπορέσει να απορροφήσει και να δεχτεί τη χώρα αυτή, την εν λόγω χώρα, εν πάση περιπτώσει. Με αυτόν τον τρόπο ε, θα εμβαθύνουμε τις δομές Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην προσπάθεια αυτή. Θα πρέπει να γίνει επίσης στο τέλος των διαπραγματεύσεων ενδεχομένως και μια δεύτερη μελέτη αντικτύπου. Ε, Μερικέ φορέ θα πρέπει βεβαίως να μπορούμε να παρεκκλίνουμε αν, ε, χρήζουν, αν υπάρχουν αποχρόντε λόγοι από τους κανόνες Ε, η ικανότητα απορρόφηση είναι βασικό θέμα και προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα της πολιτικής ε, διεύρυνσης και για τη διαδικασία ένταξης. Αλλά θα πρέπει να υπερβάλλουμε. Μέχρι στιγμής οι διευρύνσεις ε, δεν γινόταν εις βάρος της διαδικασίας ε, ολοκλήρωσης και τα διάφορα κύματα διεύρυνση συνοδεύτηκαν με μεταρρυθμίσεις των συνθήκων που επέκτηναν τις λειτουργίες και τις αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν προκλήσεις στη διεύρυνση. Μαζί με αυτές θα πρέπει να δούμε και ποια είναι τα... να μιλάμε για τα ωφέλη και για τα σημερινά κράτη-μέλη σε επίπεδο αξιών, ε, που είναι σημαντικό εργαλείο ε, δράσης ε, για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Υπάρχει θαυμάσια έκθεση της Κομισιόν του 2009, ακριβώς για αυτό το θέμα, που μίλησε για, τις, για το πώς εξελίχθη πως ήταν υποφελής η διεύρυνση για το εμπόριο, για τις επιχειρήσεις, πέντε χρόνια μετά την, το τελευταίο κύμα, το 2004 δηλαδή. Ε, και πως οι 12 νέες χώρες την έκαναν ε, πιο ισχυρό παίχτη και οικονομικά και πολιτικά. Ε, η διεύρυνση ήταν θετική και για τα παλιά και για τα καινούργια κρατημέλη. Χρειαζόμαστε, αυτό να το πούμε, στους πολίτες μας, να τους πείσουμε και να εμπλέξουμε νέους ανθρώπους, ε, να έρθουμε σε επαφή με νέους ε, ακτιβιστές, ε, δημοσιογράφους κτλ. και να τους διαμηνήσουμε αυτό το πράγμα. Το τελευταίο θέμα, οι διμερείς διενέξεις και διαφορές. Επαναλαμβάνω τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι τα διμερεί θέματα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εμπόδιο στη διαδικασία ένταξης θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με πικοδομητικό πνεύμα και το συντομότερο δυνατόν, λαμβάνοντα υπόψη τα συνολικά συμφέροντα και τι αξίε Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι θα θυμόμαστε και ξέρουμε ότι οι καλέ σχέσει γειτονία είναι βασικό κλειδί, ε, βασική προπόθεση για την ένταξη μια χώρα. Με βάση τι συνθήκε Ευρωπαϊκή Ένωση και τις, ε, τη χάρτα και τι διατάξει, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υποστηρίξει προσπάθειε για να επιληθούν ακόμα προβλήματα που υπάρχουν σε τέτοια σχέσει. Σε αυτή την προσπάθεια, αυτή η προσπάθεια μάλλον, θα είναι προ όφελο τη διεθνού επιρροή τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θα δημιουργήσει τι προποθέσει για καλύτερη συνεργασία μεταξύ των εταίρων μετά την ε, ένταξη. Για μένα, το μεγαλύτερο όφελο που μπορεί να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτέ τι διανέξει είναι το να περάσει τις ιδέε τη για συμβιβασμό, και να δείξει ότι είναι η ζωντανή απόδειξη ότι είναι δυνατόν να επιληθούν αυτά τα προβλήματα και ότι είναι επιθυμητό. Θα πρέπει να επιμείνει ότι οι διενέξεις μεταξύ γειτόνων θα πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω ε, διαλόγου, μέσω περιφερειακών λύσεων, μέσω συμβιβασμών και μέσω ε, διαρκούς προσπάθειας για συνδιαλλαγή. Τις, δια, τις ε, λεπτομέρειες της διαβάζετε στην έκθεση. Να σας πω ακόμα μια φορά ότι το να διατηρήσουμε την αξιοπιστία της διαδικασίας ε, διεύρυνσης, αυτό είναι προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια στρατηγική ανάγκη μάλιστα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς αξιοπιστία η Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύει να χάσει την ικανότητα μετασχηματισμού που έχει και την ικανότητα να επηρεάσει τις εξελίξεις ε, στην άμεση περιοχή της. Ε, θα δημιουργήσει αμφιβολίες για τη θέλησή της να κρατήσει τις υποσχέσεις της. Και αυτό σημαίνει ότι χάνει και την δύναμη που έχει και χάνει ε, ένα σημαντικό εργαλείο για την εξωτερική της δράση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να σταματήσω από εκεί που σταμάτησε η κυρία Κοπά, την αξιοπιστία της όλης διαδικασίας δηλαδή και θα ήθελα να τονίσω ότι και εμείς πιστεύουμε πάρα πολύ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η αξιοπιστία της ε, διαδικασίας διεύρυνσης θα πρέπει να διαφυλαχθεί. Αν θέλουμε να διαφυλάξουμε πραγματικά τις δυνατότητες μετασχηματισμού ε, της Ένωσης σε μια ήπια δύναμη και το γεγονός ότι δεν μπορούμε να καταφέρουμε σε μια περιοχή που είναι πραγματικά η αυλή της Ένωσης. Αν αποτύχουμε δηλαδή μπροστά στο σπίτι μας, πώς να έχουμε αξιώσεις, να έχουμε επιτυχημένη διεθνή παρουσία αλλού, σε πιο μακρινές περιοχές. Καλωσορίζουμε ε, την έκθεση της κυρίας ε, Κόπα και ιδιαίτερα ε, την μακροπροοπτική που έχει δώσει στην ίδια την έκθεσή της. Δεν θα επεκταθώ πάρα πολύ στην ουσία της έκθεσης, στο περιεχόμενο. Έχουμε κάποιες ειδικέ παρατηρήσεις τις οποίες θα διαβιβάσουμε άμεσα στην κυρία Κοπά. Αλλά η κοινωνική διάσταση την οποία τόνισε στην έκθεσή της είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν πιστεύουμε εμείς ότι χρειάζεται να προσθεθούν νέα κριτήρια στα κριτήρια της Κοπεχάγης που ήδη υπάρχουν. Ταυτόχρονα όμως πιστεύουμε ότι μπορούμε να εργαστούμε με τρόπο πιο ουσιαστικό προς δύο κατευθύνσεις. Ε, πρώτον, να δώσουμε περισσότερη ουσία και περιεχόμενο στα αντίστοιχα κεφάλαια ε, κατά τη διαδικασία διαπραγματεύσεων και εδώ σκέφτομαι ιδιαίτερα το κεφάλαιο 19 για τις κοινωνικές πολιτικές, αλλά και με πιο στοχευμένη βοήθεια έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι οι χώρες αυτές της διαδικασίας διεύρυνσης θα μπορέσουν να βελτιώσουν τις κοινωνικο-οικονομικές τους ε, ε, συνθήκες κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης πιστεύουμε ότι είναι σημαντική η προσέγγιση με τη συγκριτική αξιολόγηση, τα ορόσημα, τα benchmarks, για να υπάρχει και ε, διαφάνεια και δικαιοσύνη στη διαδικασία. Να βεβαιωθούμε ότι δεν δημιουργούνται έτσι προσκόμματα και αντιπέρβλητα εμπόδια για κάποιες χώρες, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο τονίζει και η ίδια η κυρία τα είπε προηγουμένως στην εισαγωγή της. Θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να θέσουμε προτεραιότητες στις προσπάθειες, στις πολιτικές που θα έχουμε το διαπραγματευτικό μας πλαίσιο και όπως είπαμε να λάβουμε υπόψη ιδιαίτερα τη διάσταση του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών ελευθεριών. είναι ένα συστημικό στοιχείο που θα πρέπει να ε, αποτελεί το θεμέλιο όλων των διαπραγματεύσεων ε, προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιτρέψτε μου, Πρόεδρε, να αφαιρθώ δύο λεπτά σε ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να σας ε, αναφέρω. Σήμερα το πρωί Επιτροπή ενέκρινε την έκθεση παρακολούθησης για τη προετοιμασία ένταξης της Κροατίας. Όπως μπορεί να θυμάστε, ε, είναι μια τακτική διαδικασία που προβλέπεται στη συμφωνία στη συνθήκη προσχώρησης της ε, Κροατίας και είναι μάλιστα η πρώτη έκθεση μετά την υπογραφή της συνθήκης. Ε, αξιολογείται η πρόοδος που έχει καταβάλει η Κροατία κατά το εξάμεινο Σεπτεμβρίου 2011 με Φεβρουάριο 2012 και εστιάζει κυρίως σε τρεις ε, τομείς. Ε, ανταγωνισμός, ε, δικαιοσύνη, ελευθερία ασφάλεια και δικαστικό σύστημα. Η Κροατία προοδεύει στο δρόμο της ένταξης και είναι πεπισμένη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η Κροατία θα κάνει όλα τα τελευταία βήματα που χρειάζεται έτσι ώστε η χώρα είναι πλήρως έτοιμη για να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Ιουλίου του 2013. Παραμένουμε προσιλωμένοι στην κατεύθυνση αυτή και στην εξασφάλιση της επιτυχούς ένταξης της Κροατίας και θα εξακολουθήσουμε να παρακολουθούμε ε, πολύ στενά τις εξελίξεις και τι θα κάνει η Κροατία, πώς θα ανταποκριθεί στις ε, υποχρεώσεις που ανέλαβε, έτσι ώστε να είναι ομαλή η ένταξή της και είναι ε, κοινό μέλημα και στόχος και της Ένωσης και της Κροατίας αυτό. Τα τονίζω αυτά τα στοιχεία διότι έχω την αίσθηση ότι εντάσσεται αυτό και στην έκθεση της κυρίας Κοπά. Δηλαδή να δώσουμε μια νέα όθηση στη διαδικασία της διεύρυνσης και με τη δική σας βοήθεια και υποστήριξη θα είμαστε σίγουρα σε θέση να υπερβούμε την κόπωση που ανέφερε η κυρία Κοπά. Και ε, ξέρετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είναι ταμπού αυτή η λέξη, αλλά δεν θέλω να επεκτάθω σε αυτό. Είναι Ε, κοινό μας ενδιαφέρον να συνεχιστεί με αξιόπιστο τρόπο η διαδικασία της διεύρυνσης, να υπάρχει μετασχηματισμός ε, και ε, πρόοδος και μετάβαση στα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων. Ευχαριστώ πολύ. Ο ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση αυτή. Για τη σημερινή απόφαση και τη θέση σας για την έκθεση. Τώρα έχουμε πολλούς εγγεγραμμένους ομιλητές. Ερωτήσεις φαντάζομαι. Πόσο χρόνο έχουμε για αυτή τη συζήτηση. 20 λεπτά. Οι σκιώδεις συζητητές 2 λεπτά και οι υπόλοιποι 1 λεπτό για να προκάνουμε. Η κυρία Όμεν Ρόιτεν. Ναι, πρόεδρε. Θα προσπαθήσω. Τι να κάνω. Ευχαριστώ. Ε, συμφωνώ, πρόεδρε, με την κυρία Κοπά ότι η διεύρυνση είναι σημαντική απάντηση στη διπλή πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, η εδραίωση του δικού μας ρόλου στον κόσμο και η σταθεροποίηση του άμεσου περιβάλλοντός μας. Ε, πρόεδρε, η διαδικασία διεύρυνση είναι και παραμένει σημαντικό εργαλείο προ την κατεύθυνση αυτή. Αλλά θα πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί, γιατί δεν είναι αυτό σκοπό η διεύρυνση. Είναι μέσον. Είναι μέσον για να φτάσουμε σε κάποιου στόχου μα. Και αυτό σημαίνει επίση να δούμε και τη δυνατότητα ενσωμάτωσης της ε, Ένωσης κάποιων νέων χωρών. Ευχαριστώ την κυρία Κοπά για όλα αυτά που έχει γράψει, αλλά διερωτώ με πρώτον αν η έκθεση αυτή και οι συστάσεις ε, έχουν περισσότερη δύναμη και περισσότερο σθένος όταν είναι πιο, αν είναι πιο σύντομη η έκθεση γιατί νομίζω ότι είναι πολύ αναλυτικά και οι αναφορές σε πολλά πράγματα δεν θα πρέπει να είναι επανάληψη των όσων λέμε για τις διάφορες χώρες η έκθεση αυτή επίσης δεν θα πρέπει να προτρέχουμε πάρα πολύ όταν μιλούμε για την προταξιακή ε, στήριξη και κάτι άλλο που μου λείπει από την έκθεση είναι το εξής λέτε τα υποψήφια κράτη και τα ενδεχομένα υποψήφια ε, έχουν την αίσθηση ή τους δίνουμε την αίσθηση ότι μπορούν να μπουν στην Ένωση. Αλλά για την εισηγήτριά μας, πού είναι τα γεωγραφικά σύνορα της Ένωσης. Και για τα διμερή θέματα επίσης. διμερή ε, Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Διαρωτώ με. Τι γίνεται με τα διμερή αν υπάρχουν διμερεί θέματα πριν να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις ή μήπως πρέπει να έχουν λυθεί αυτά πριν αρχίσουν διαπραγματεύσεις. Τώρα τη συμπληρωματική ε, χρηματοδοτική ενίσχυση για τα κοινωνικά θέματα στις υποψήφιες χώρες. Ε, η, ε, η πολιτική επικοινωνίας. Ζητείτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βρουν νέα μέσα για κάποια άλλα κριτήρια κοινωνικά ενδιαφέροντα είναι, αλλά πώς θα σταθμιστούν. Κοιτά τους παραγράφους 3, 5 και 6. Θα πρέπει να δούμε την πρόοδο και να ε, την αξιολογήσουμε. Και ένα σύστημα παρακολούθησης να υπάρχει και αξιολόγησης και ε, ελέγχου των χωρών. Λοιπόν, όταν τα ζητάμε όλα αυτά, πού είναι το καθαρό μήνυμα που πρέπει να στείλουμε. Μήπως χάνεται λίγο μέσα σε όλο αυτό τον όγκο των ε, προτάσεών μας. Επί της ουσίας δεν διαφωνούμε, αλλά για να λειτουργούμε αποτελεσματικά θα πρέπει να έχουμε ένα μήνυμα ε, πιο ισχυρό, πιο καθαρό και να μην χάνεται μέσα σε όλο αυτό τον όγκο των προτάσεων. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Chair. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Πιστεύω ότι όντω πρόκειται για μια εξαιρετική έκθεση. Ευχαριστώ την κυρία Κοπά. Και είναι πολύ κοντά στη δική μου άποψη περί διεύρυνσης. Χαίρομαι διότι στην αιτιολογική σκέψη F λέει ότι κάθε χώρα θα πρέπει να κρυφεί βάσει των δικών της επιτευγμάτων. Και βεβαίως ε, θα πρέπει να υπάρχουν ε, για όλους ταυτόσιμα κριτήρια και θα πρέπει ό,τι γίνει να γίνει με διαφανή τρόπο. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει τελικά να κάνουμε κάτι το, αν θέλετε, μια τεχνική αξιολόγηση προοδεύοντας ε, έχουν τηρηθεί τα κριτήρια, έχουν, ε, πληρούνται, προχωρήστε στο επόμενο βήμα. Αυτό το Σαββατοκύριακο, όπως ξέρετε, παρετήθηκε η δική μας κυβέρνηση Ολλανδική, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα υπάρχουν πληρωματικές δυσκολίες για τους Ολλανδούς. Και ίσως αυτό οδηγήσει στο να επιτευχθούν κάποιες συμφωνίες πιο εύκολα στο επίπεδο Συμβουλίου. Τώρα, για τα θέματα τα διμερεί. Εμένα με ικανοποιούν τα άρθρα 11 και 12 στην εκθεσή σας. Και μία παρατήρηση για την κοινωνική διάσταση. Σήμερα στην Επιτροπή Επασχόλησης εγκρίναμε γνωμοδότηση για το... Uh, Είπα δύο και αυτό ίσως έχει σχέση με τα, τι μπορεί να γίνει πρώην και ίσως έχει σχέση αυτό με τα κοινωνικά κριτήρια. Οι στόχοι για την Ευρώπη του 2020 συνάδουν και με την εκεί και με την ε, οικονομική ανάπτυξη και ίσως θα πρέπει να κάνουν το ίδιο και οι χώρες υποψήφιες ώστε να ευθυγραμμιστούν σιγά ώστε να μπορέσουν να συμπεριληφθούν στην ε, φόρο αυτή και ευρωπαϊκή οικονομία στην οποία θέλουμε, από την οποία θέλουν να αποκλείεται κανείς. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δαφ, πρόεδρε. Πρόκειται για μια έκθεση με πολλές προκλήσεις. Πριν όμως να αναφερθούμε στα κριτήρια της Κομπεχάης θα πρέπει να αναρωτηθούμε για ποιο λόγο θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Βάσει της σημερινής μας εμπειρίας, τι πήγε στραβά σε θέματα διεύρυνσης και περαιτέρω και θα πρέπει να... Κάποια κράτη-μέλη, εάν αρχίσουμε να πηγαίνουμε πολύ μακριά στο θέμα αυτό, να αναθεωρήσουν και το δική τους την όλη την πολιτική σε θέματα κριτηρίων. Πιστεύω ότι είναι επίσης το θέμα της αξιολόγησης τεχνικό θέμα και δεν μπορούμε να πώς τυκοποιήσουμε κάποια πράγματα, όπως πιστεύει η κυρία Κοπα. Πρόκειται για μια βαθιά πολιτική διαδικασία. Και αν εμείς δεν υλοποιήσουμε τις υποσχέσεις μας, προς κάθε κατεύθυνση, η ίδια η Ευρώπη θα υποστεί πλήγμα στην ε, πολιτική δύναμη που θέλει να έχει στην παγκόσμια κοινωνία που ζούμε σήμερα. Υπάρχει και η ηθική διάστηση Και θα πρέπει να κρατήσουμε το λόγο μας όσον αφορά την διεύθυνση σε σχέση με τους ενδυνάμει υποψηφίους. Τώρα, όσον αφορά την οικονομική και κοινωνική πολιτική, δεν θα πρέπει να υποτιμήσουμε την μεγάλη, τις μεγάλες αποκλίσεις που υπάρχουν επί συνταξή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας υπάλληλο στο Βέλγιο κοστίζει έναν ώρα 35 ευρώ. Ενώ σε μια άλλη χώρα μπορεί να κοστίσει αυτό στον εργοδότη 2,5 ευρώ. Η κοινωνική διάσταση είναι ένα θέμα, το κοινωνικό dumping είναι ένα άλλο όμως. Και τελικά πιστεύω ότι θα πρέπει να μελετήσουμε πιο λεπτομεριακά τις προτάσεις που συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση αυτή. Γιατί αν θέλουμε να αλλάξουμε όλη τη διαδικασία προσχώρησης, εμείς ως ομάδα θα θέλαμε να τονιστεί πολύ περισσότερο το άνοιγμα των κεφαλαίων 23 και 24 στην αρχή της όλης διαδικασίας διαβρύνσης. Αυτό το υπαγορεύει η εμπειρία μας με την Τουρκία και με την Κροατία. Ίσως όσο προχωρούμε προς το 2015 θα πρέπει να μπορέσουμε να προωθήσουμε και την ιδέα του συνδεδεμένου κράτους. Που ίσως να είναι η καλύτερη δυνατή λύση για κάποιες ενδυνάμει υποψήφιες χώρες. Παρακαλώ να μην ξεπερνάτε ο καθένας τον χρόνο που έχετε διότι έχουμε ακόμη την έκθεση Λάμπστορφ και τον εκπρόσωπο της UNESCO και στις 5.30. Όταν λοιπόν θα έχουμε να εξετάσουμε την έκθεση αυτή με τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί από τους συναδέλφους, θα αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο και θα έχουμε την δυνατότητα να μπούμε σε περισσότερε λεπτομέρειε. Ο κύριο Κατσίν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ την κυρία Κοπά για την εξαιρετική έκθεσή τη, στην οποία τονίζονται όλα τα κύρια θέματα για μια επιτυχή διαδικασία προσχώρηση. Μία από τι προ... Ε, τις τροπολογίες που θα καταθέσω έχει να κάνει με τον ρόλο τη επιτροπή. Δεδομένου ότι, στη, κάποιοι, ότι πάλι της ευρωπαϊκή Ένωσης μεγάλου σεβασμού σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θα πρέπει να ζητήσουμε λοιπόν από την Κομισιό να, ε, ε, ενεργήσει αν θέλετε ε, με πιο δυναμικό τρόμα, τρόπο για θέματα τα οποία αφορούν σε κάθε χώρα θέματα που είναι πολύ δυνατά. Θα πρέπει λοιπόν ο καθένας να μπορεί κυρίω για κάθε χώρα να μας δίνει συγκεκριμένα παραδείγματα σε θέματα διαφθοράς και δωροδοκίες. Δεν κάνει τίποτε ε, το ειδικό, όλα είναι γενικά. Αυτό που λέγει η Επιτροπή ότι ε, στην αρχή του διαπραγματεύσεων προτίθεται να ανοίξει τα κεφάλαια 23-24 θα επιταχύνει την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι δεν επαρκεί αυτό. Πολλά περισσότερα πράγματα μπορούμε να κάνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Που έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ε, και με ένα όραμα για το μέλλον και όχι μόνο στις λεπτομέρειες. Τι θα πούμε στους νέους που γεννήθηκαν το 90 και τώρα ρωτάνε τι μέλη γενέστε, τι μπορούμε να κάνουμε, πώς θα προχωρήσουμε. Γιατί άκουσα την κυρία Όμεν Ρόιτεν. Και τι είναι αυτή η αμυντική στάση. Ε, είναι σαν να μην θέλετε καθόλου διεύρυνση που λέτε ε, ότι δεν είναι αυτός σκοπός. Και ποιος είναι ο σκοπός και πώς μπορούμε να αποφασίσουμε, γιατί σε 20 χρόνια μπορεί να είναι τελείως διαφορετική η ε, κατάσταση από ότι το 1985. Αν το 1985 είχαμε αποφασίσει για πώς θα έχει η Ευρώπη οριστικά, δεν θα κάναμε καμία διεύρυνση. Και πώς μπορεί κανείς να ανέχεται κυβέρνηση... Ε, την κυβέρνηση του κύριου κύριος που είναι τα πάντα εκτός από φίλους της Ευρώπης. Πολλές τροπολογίες θα έρθουν για να καταλάβουμε ποιο θέλει τη διεύρυνση στο Κοινοβούλιο και με ποιου όρου και προποθέσει. Και χαίρομαι και για τη δήλωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και στο πρόσωπο του Επιτρόπου Φίλου έχουμε ένα επίτροπο οραματιστή που να σκέφτεται και το μέλλον. Για να φύγουμε ε, από το σπιτάκι μα ο καθένα, να κοιτάξουμε και πέρα από το φράχτη, να ανοίξουμε. Μα δεν χρειαζόμαστε ένα Βίλντερς, έχουν τους σοσιαλδημοκράτες, αν μπαίναν στην κυβέρνηση αυτή δεν θα τον είχαν ανάγκη το Βίλντερς, λέει ο πρόεδρος. Ο κύριος Κούκαν. Äh, λοιπόν, κύριε Κράιζελ Ντόφλερ, αν θέλετε να το δείτε κομματικά και με τις χώρες, να δούμε τι γίνεται στις κάτω χώρες και τι κάνουν σοσιαλδημοκράτες του κόμματο τη ε, εργασία, του ΠΒΔΑ, ότι νύπτουν τα σχήρα του και δεν αναβάνουν κυβερνητικέ ευθύνε. Έχει σχέση και αυτό με αυτά που λέμε, έτσι. Δυστυχώ αυτό είναι το πρόβλημα όλο και περισσότερο έχουμε ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη και όχι αρκετά δημοκρατικά που να θέλουν να συνασπίζονται και να κάνουν ε, πλειοψηφίες και εξαρτώμαστε από τέτοια ακροδεξιά από κόμματα και είναι τεράστιο το πρόβλημα, πιστέψτε με. Ο κύριος Κούκαν. Ευχαριστώ. Η δουλειά και τα αποτελέσματα της κυρίας Κοπά νομίζω ότι θα πρέπει να τα εκτιμήσουμε. Στην περίπτωση των Δυτικών Βαλκανίων. Μην ξεχνάμε την μετασχηματιστή ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ένωση και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί πιο αποτελεσματικά. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε και την οικονομική και κοινωνική διάσταση, που είναι σημαντικός παράγοντας, αλλά δεν θα πρέπει να υπερτονίσουμε τη σημασία τους. Η Κομισιόν προσπάθησε Σχάτως να δείξει καινοτόμο πνεύμα στην, στον τρόπο που προσεγγίζει τη διαδικασία διεύρυνσης. Θα πρέπει να την εκτιμήσουμε αυτή την προσπάθεια, θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις πρωτοβουλίες της και εμείς θα πρέπει να είμαστε και πιο ευέλικτοι στο κάτω-κάτω προς αυτή τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Σε περιπτώσεις, δηλαδή εννοώ, που δεν μπορούν να θεωρηθούν κλασικές, όπως το Κωσφοπέδιο ή η Βοσνία Ζεγοβίνη. Επίσης, θα πρέπει να αφιερώσουμε περισσότερο χώρο σε αυτή τη διαδικασία στο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί συχνά μπορούμε να συνεισφέρουμε και εμεί την όλη διαδικασία και να βοηθήσουμε να γίνουν κάποιες πολιτικές εξελίξεις. Έχουμε μοναδική πολιτική εμπειρία ε, με πολλούς ευρωβουλευτές από τις νέες χώρες που με κάποιο τρόπο είχαν ήδη εμπλακεί στη διαδικασία ολοκλήρωσης ε, και διεύρυνση και νομίζω ότι την πείρα των ανθρώπων αυτών θα πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε. Ευχαριστώ. Γκόμε, Ευχαριστώ την Ελένη Κοπά για την έκθεση και τα ενδιαφέροντα στοιχεία που εμπεριέχει η έκθεσή της. Υποστηρίζω την έκκληση για τα κοινωνικά πρότυπα που θα πρέπει να τα προτάξουμε στην αξιολόγηση της ε, διαδικασίας της ε, διεύρυνσης. Ο λόγος που τα κοινωνικά πρότυπα δεν θα είναι τόσο πολύ, δεν είναι τόσο σημαντικά, είναι ότι τα έχουμε υποτιμήσει και εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, τα αποδομούμε αυτά τα κοινωνικά πρότυπα εμείς εδώ. ας πούμε, η διαδικασία μεταρρυθμίσεων στη χώρα μου, αυτό σημαίνει η αποδόμηση των κοινωνικών προτύπων ε, στη χώρα από την Πορτογαλία. Ε, επομένως, τα κοινωνικά πρότυπα και για τις υποψήφιες χώρες, αλλά και για μας, ε, θα, θα πρέπει να τα λαμβάνουμε περισσότερο υπόψη μας. Επίσης, ε, ένας μηχανισμός παρακολούθησης, το υποστηρίζω, για να δούμε πώ θα εφαρμόζονται τα κριτήρια τη Κοπενχάγη, όχι μόνο στι υποψήφίε χώρε, αλλά και στι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δεν μπορούμε να είμαστε αξιόπιστοι και να υλοποιήσουμε του ε, στόχου που υποτίθεται θέλουμε να υλοποιήσουμε, ε, τη στιγμή, όταν τη στιγμή που ζητάμε από τι υποψήφιε χώρε κάποια πράγματα, εμεί τα ξεχνάμε εντελώ αυτά τα πρότυπα, τα παραβλέπουμε. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις ε, που αποδεικνύουν αυτό που λέω. Δεν συζητάω καν το θέμα της ε, ε, συνεργασίας κάποιων χωρών με τις ε, πτήσεις αυτές που οδήγησαν σε βασανιστήρια. Τα κοινωνικά πρότυπα έχουν τόσες επιπτώσεις για τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, τις ελευθερίες κτλ. Ο κοινωνικός διάλογος, η ελευθερία των συνδικάτων κτλ. Τέλος, εκφράζω την ανησυχία μου για τα το θέμα των διμερών διενέξεων. Παραδείγματο χάρη, η διμερή διαφωνία Κύπρου και Τουρκία μπορεί να μα δημιουργήσει εμά προβλήματα το επόμενο εξάμεινο. Ε, της, δεδομένων των πολύ προκλητικών σχολείων των τουρκικών αρχών. Ελπίζω να συνειδητοποιούν ότι με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο ενοχλούν την Κύπρο, αλλά την Ευρωπαϊκή Ένωση την ίδια ενοχλούν. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει τίποτα προκλητικό σε αυτή την έκθεση. Δεν καταλαβαίνω πού είδε αυτές προκλήσεις ο κύριος Νταφ. Είναι μια καλή απόπειρα, νομίζω, να προσπαθήσουμε να σκεφτούμε τα αποτελέσματα της διεύρυνσης και τις ε, προοπτικές που έχουμε για τις μελλοντικέ διευρύνσεις. Προσπαθούμε να ξεχωρίσουμε τη διαδικασία από τις συγκεκριμένες χώρες που εξετάζουμε, που έχουμε απέναντί μας ε, σε αυτή την ε, διαδικασία διεύρυνση. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή συνεισφορά η έκθεση αυτή, ακριβώ για τους λόγους που προανέφερα, και πιστεύω ότι θα δώσει αποτελέσματα και θα καταστήσει τη δική μα προσέγγιση απέναντι στη διεύρυνση και πιο σοφή και πιο αξιόπιστη. Κάποια θέματα τώρα που θέλω, να να σταθώ. Καταρχά είμαι λίγο σκεπτικιστή για αυτή την ιδέα προσμέτρησης του δυναμικού α, ένταξη. Γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθεί από αυτού που είναι κατά τη διεύρυνση για να αποδεικνύουν συνέχεια ότι δεν υπάρχει πιο δυναμικό. Και τελικά να βλάψουν την όλη διαδικασία. Κάτι που δεν θα θέλαμε. Δεύτερον, την παρακολούθηση των κριτηρίων ε, ένταξης. Είμαι υπέρ της ιδέας να έχουμε ένα μηχανισμό παρακολούθησης για όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο για τις υποψήφιες χώρες για αυτούς που έχουν προσχωρήσει πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ακόμα και τώρα μπορούμε να δούμε τουλάχιστον τρεις χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ίσως να μην πληρούν πλήρως αυτά τα κριτήρια. Και τέλος, αυτή την έκθεση θα πρέπει να αναφέρουμε ότι και οι χώρες διεύρυνσης και οι υποψήφιε χώρε δηλαδή θα πρέπει να σέβονται τι στρατηγικέ μα. Παραδείγματο χάρη την ε, στρατηγική Ευρώπη 2020. Ε, ξέρω ότι στην οικονομική κατάσταση που βρισκόμαστε ε, είναι λίγο δύσκολο να μιλάμε για αυτή τη στρατηγική, αλλά κάπου πρέπει να βάλουμε και αυτή την, ε, αυτό τον χρονικό όριζο του 2020. Τέλο, θέλω να πω ότι είναι μια θαυμάσια προσπάθεια. Θυμάμαι τι συζητήσει που έγιναν στο Διευρυμένο Προεδρείο όταν αποφασίζαμε για την έκθεση αυτή, ότι ίσω ε, να είναι επικίνδυνη μια τέτοια έκθεση. Ε, μπορεί να μην ξέρουμε πού θα καταλήξει, αλλά το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ήταν πάντα υπέρ των διευρύνσεων. Και το θέμα είναι πώ μπορούμε να καταστήσουμε τη διαδικασία πιο αξιόπιστη. Και να μην χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκθεση ω αφορμή για να μπλοκάρουμε τι διευρύνσει. Ε, μην ξεχνάμε ότι είναι μία από τι ε, βασικέ ε, πολιτικέ Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόεδρε, ο κύριος Στάνοφ, είναι η έκθεση της ε, ε, καλή, αλλά δεν συμφωνώ με ένα μοντέλο ε, για όλου, κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σαν το ευρώ να μπουν, α πούμε, όλε οι υποψήφιες χώρες στο ευρώ. Αυτό θα ήταν όλεθρο. Μπορεί να είναι τεχνική διαδικασία, κάποιο είπε, αλλά χρειάζεται πολιτική συμφωνία και σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου. Και γεωγραφικά πώ ορίζεται η Ευρώπη, η πολιτικά. Μέχρι πού φτάνει. Και αυτό χρειάζεται και δημοκρατική υποστήριξη από τους ψηφοφόρους μας που θα πρέπει να δεχθούν ε, το ενδεχόμενο κόστος για τους φορολογούμενους, τα διαρθρωτικά ταμεία, την ΚΑΠ και άλλες επιδοτήσεις. Και μπορεί να έχουμε και πολύ μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών και αυτό επιβαρύνει τους δημόσιους προϋπολογισμούς. Είδαμε το 20% ψήφισε στη Γαλλία την κυρία Λεπέν. Και προσωπικά πάντα ε, ήμουν ε, κατά, ε, του, είχα λυπηθεί που δεν δώσαμε καθεστώς ενδεχόμενης υποψήφιας χώρα στην Ουκρανία. Και έχουμε την Αλβανία, ας πούμε, ενδεχόμενη υποψήφια χώρα. Υποστηρίζω και εγώ την παραγραφό 12, αλλά θα ήθελα να συμφωνήσουν με συνθήκη όλες οι χώρες να μην χρησιμοποιήσουν διμερείς διενέξεις για ονόματα, για ε, εσωτερικά εκτοπισμένους ε, για σύνορα για να μπλοκάρουν πράγματα με διάφορες ε, γειτονικές χώρες όπως είδαμε με τη Μακεδονία ας πούμε ή με την Κροατία που Ελπίζω ποτέ να με χρησιμοποιήσει το νέο καθεστώ για να μπλοκάρει την είσοδο τη Σερβία για κάτι που έγινε πριν από 10 και πλέον χρόνια. Και αυτό που είπε ο κύριο Κούνκαν, ενδιαφέρον. Ακόμα και πριν τη συνθήκη τη Λισαβόνα, το Κοινοβούλιο, ε, μοναδικό είναι αυτό, είχε περισσότερε εξουσίε στη σύμφωνη γνώμη ε, για μεμονωμένε χώρε. Και τη συμπερασμένη ε, διεύρυνση που γίναμε από 15-25 ε, σε σχέση με τα εθνικά κοινοβούλια που δεν μπορούσαν να βάλουν βέτο για μεμονωμένες χώρες. Δηλαδή από πλευρά της συνθήκης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει περισσότερες εξουσίες από τα εθνικά κοινοβούλια και καλό θα ήταν να το αξιοποιήσουμε προς το δικό μας συμφέρον και για να αυξηθεί και η επιρροή μας στην όλη διαδικασία και διεύρυνση. Ευχαριστώ. Ποιος άλλος είχε το λόγο. Α, ο κύριος Σόλτς είχε ζητήσει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ είμαι σκιώδη ηγητής και μου δίνετε το λόγο. Θυμάστε τις ε, εκθέσεις το 2006 και το 2008 για αυτό το θέμα και καλό είναι να θυμηθούμε καταρχήν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανοιχτή για όποιον θέλει να ενταχθεί στην Ένωση, για όλες τις χώρες. Και αυτό το ξαναβλέπω στην έκθεση ε, της κυρίας Κοπά και θέλω να την ευχαριστήσω ιδιαίτερα ε, για τη ε, ισχυρή της δέσμευση και το σθένος της προς την κατεύθυνση αυτή. Το 17 το θεωρώ πολύ σημαντικό. Ακόμα και αν τα συζητούμε θα πρέπει να εφαρμοστεί σε πρακτική πολιτική αυτό το δικαίωμα και να συμμετέχουν και οι πολίτες μας. Όταν μιλούμε για τη διεύρυνση, να συμμετέχουν, ιδιαίτερα στην παρούσα φάση και την ιδιαίτερη εξέλιξη στο ιστορικό της Ένωσης. Γι' αυτό η δυνατότητα απορρόφησης και ενσωμάτωσης νέων χωρών είναι σημαντική και είναι και πρόκληση όταν συζητούμε και για τη διεύρυνση γενικότερα και ε, μας απασχολεί αυτό το θέμα. και θα πρέπει να έχουμε και μια εσωτερική συνοχή 27-28. Ε, ποια είναι τα κοινωνικο-οικονομικά θέματα και η συνοχή. Και αυτό τα γράφει η έκθεση και την κοινωνική διάσταση, πάρα πολύ σημαντικό. Δύο λόγια μόνο για τα κριτήρια της Κοπενχάγης. Νομίζω θα πρέπει να τα τηρήσουμε, να τα διατηρήσουμε και να σκεφτούμε πώς μπορούν να μετεξελιχθούν, αλλά και σοβαρά να ασχοληθούμε και τα 27 κράτη και να πούμε Άραγε σήμερα θα μπορούσαμε να είχαμε συμφωνήσει σε αυτά τα κριτήρια. Αυτό που συμβαίνει στην Ολλανδία, στην Ουγγαρία και αλλού. Τι γίνεται με τις πολιτικές ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα στην ίδια την Ένωση και ζητούμε από άλλες χώρες ε, αν θέλουν να ενταχθούν να τα πληρούν. Θα πρέπει και ε, στο μέλλον αυτά τα θέματα να μας απασχολήσουν. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να κάνω και εγώ μερικές παρατηρήσεις, λέει ο Πρόεδρος. Δεν λέει συνθήκη ότι μπορεί οποιαδήποτε χώρα ε, να μπει. Όποια χώρα πληρεί τα κριτήρια και είναι ευρωπαϊκή μπορεί να κάνει αίτηση για ένταξη. Ε, μικρή διαφορά. Δεν είναι αυτόματο ότι άμα κάνεις την ένταξη θα μπει κιόλα. Είναι σημαντικές ε, κάποιες προτάσεις κυρία Σκοπά. Αυτό με το post-monitoring. Θα πρέπει να το σκεφτούμε πολύ ε, για να κερδίσουμε και τον πληθυσμό και τον κόσμο στο πλευρό μας. Στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία το είδαμε και ε, με άλλη ευκαιρία, αλλά δεν λειτουργήσε ποτέ. Και θα πρέπει να σκεφτούμε γιατί έλειπε και το πολιτικό θάρρος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιοποιήσουν αυτό το μηχανισμό. Και θα πρέπει να συζητήσουμε και μεθόδους κάποια στιγμή για να έχουμε μια αξιόπιστη υπόθεση. Διότι είναι σημαντικό κάτι τέτοιο για να ε, δώσουμε και κάποια ασφάλεια στους ίδιους τους λαούς μας και να διευκολύνουμε τις διευρύνσεις. Επίσης θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλάβουμε και να δεχτούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πολίτες έχουν κάνει τεράστιες προσπάθειες. Όταν έγινα εγώ Ευρωβουλευτής ήμασταν 9 κρατημέλη και τώρα φτάνουμε τα 28. Από το 2004 μέχρι φέτος έχουμε 13 νέες χώρες. Αυτό το θεωρώ τεράστιο επίτευγμα. Και γι' αυτό η διεύρυνση είναι από τις πιο επιτυχείς για πιο ή επιτυχέστερη. Αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι θα πρέπει να λειτουργεί σωστά και να εφαρμόζεται σωστά. Έχουμε και φάσεις εδραίωσης μετά τις διευρύσεις και τώρα ζούμε και περίοδους κρίσης. Και στην κρίση, το βλέπουμε και από τα εκλογικά αποτελέσματα, οι λαϊκιστές έχουν πάντα την ευκαιρία να εκμεταλλεύονται την κρίση εις βάρος άλλων. Την κρίση πάντα την εκμεταλλεύονται λαϊκιστές, δεξιοί, αριστεροί, κατά των ξένων, των μεταναστών, των διαφορετικών. Φταίνε όλοι αυτοί. Έχουμε την παλιά ιστορία. Δεν είναι σημερινή, είναι ανέκαθεν και τα ξαναζούμε αυτά τα πράγματα τώρα. Ε, αν δεν το καταλάβουμε αυτό ε, και δεν το δεχτούμε, έχουμε πρόβλημα. Και θα πρέπει με τρόπο λογικό να συζητήσουμε και σε σχέση με τη διεύρυνση πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα. Γιατί να βάλουμε το κεφάλι κάτω και να προχωρούμε δεν είναι και αυτό λύση. Θα πρέπει να μας ακολουθεί και η βάση. Εξού λοιπόν και η δυνατότητα απορρόφησης της Ένωσης και διεύρυνσης. Το είπε και η κυρία Κοπά. Είναι σημαντικό το σημείο αυτό. Η κυρία Όμεν το είπε λίγο οξύτερα. Αλλά αυτό που είπα και εγώ προηγουμένως έχει να κάνει αυτό και είναι σαφές. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να το εξηγούμε στους πολίτες και με τρόπο πιο ακριβή και πιο συγκεκριμένο. Πότε ανατρέπεται αυτή η κατάσταση κάποια στιγμή να μην είναι ε, σε θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργεί. Το πρωτογενές δίκαιο. Όταν έχουμε 35-38 κράτη, πώς αλλάζεις με ομοφωνία τις συνθήκες, για να μην πω και σε άλλους τομείς που χρειάζεται ομοφωνία. Ανέκαθεν λέγαμε ότι η συνθήκη της Λισαβόνας ήταν απάντηση για τη διεύρυνση προς τους 12 και ότι χρειάζεται ενίσχυση περισσότερο η Ένωση αν θέλουμε να προχωρήσουμε κι άλλο. Από την άλλη, έχουμε υποσχέσεις που μας υποχρεώνουν. Ε, το 2003 στη Θεσσαλονίκη υποσχεθήκαμε στα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων. Όλα αυτά θα πρέπει να συνδυαστούν. Δηλαδή οι χώρες να πληρούν μεν τις προϋποθέσεις, χωρίς εκπτώσεις βέβαια, αλλά θα πρέπει και εμείς να εργαστούμε προς την κατεύθυνση αυτή, αν θέλουμε να διευρυνθούμε, να αλλάξουν οι δομές μας για να δεχτούμε τις χώρες αυτές. Και συμπεριλαμβανωμένο εδώ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Και αυτό θα πρέπει να το δούμε, είναι συναφή αυτά τα δύο, αν θέλουμε να πετύχει η διεύρυνση. Και πιστεύω ότι η έκθεση της Σκοπά Κοπά αποτελεί καλή βάση προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά στις τροπολογίες θα πρέπει να κοιτάξουμε Μήπως πρέπει να το πούμε με τρόπο πιο έντονο για τη διαδικασία. Μετά τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, και παράδειγμα άλλο η Κροατία, κοιτάξαμε περισσότερο τη δικαιοσύνη, τη διαφθορά κτλ. Ορισμένα τα ανέφεραν προηγουμένως. Αυτά είναι καρκινώματα που εμποδίζουν τις χώρες να αναπτυχθούν. Εδώ θα πρέπει να γίνουμε πιο έντονοι και πιο οξύ στη διατύπωση για να υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας και προόδου της διαδικασίας. Και επίση θα πρέπει να πούμε και τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να δεχτεί όλε αυτέ τι χώρε, κύριε Κοπά, και να προσθέσουμε ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και στις χώρες αυτές ότι όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις που κάνουν θα έπρεπε να τις κάνουν έτσι κι αλλιώς. Μπουν δεν μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν τις κάνουν για την Ένωση. Τις κάνουν γιατί είναι η μοναδική τους ευκαιρία να προχωρήσουν και να έχουν ένα κράτος επιτυχημένο, οικονομικό, κοινωνικό και να είναι και κράτος δικαίου και δημοκρατία. Είναι γενικά προϋπόθεση. Ε, ακόμα κι αν ένα κράτος παραμένει μόνο του στη διεθνή κοινότητα. Δεν τα κάνετε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τον εαυτό σας τα κάνετε όλα αυτά. Γι' αυτό θα πρέπει να τους το πούμε και να το συζητήσουμε γιατί πολλές φορές το έχουμε ε, παραμελήσει και από τις κυβερνήσεις. Γιατί και οι κυβερνήσει του βγαίνουν και λένε και εγώ δεν συμφωνώ, αλλά κάτι ε, ηλίθιοι εκεί στις Βρυξέλλες μας τα επιβάλλουν. Όχι, πρέπει να το συζητήσουμε σοβαρά και εντατικά και στην παρούσα φάση ακόμα περισσότερο. Μήπως θα πρέπει να κάνουμε κάποιες τροπολογίες προς την κατεύθυνση αυτή. Να καλέσουμε και εμπειρογνώμονες, όχι μόνο με τις τροπολογίες. Αν θέλετε και ακρόαση να κάνουμε. Το θεωρώ τόσο σημαντικό, τόσο θέμα αρχής που δεν θα πρέπει να το διεκπαιρεώσουμε έτσι ε, διοικητικά μέσω τροπολογιών. Να το συζητήσουμε πιο πολύ. Κυρία Κοπά, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τη συνεισφορά τους, τα σχόλιά τους. Όπως κατανοείτε δεν είναι εύκολο το εγχείρημα. Αυτό το οποίο με απασχόλησε κυρίως είναι να στείλω ένα ηχηρό μήνυμα για την αξιοπιστία της διαδικασίας διεύρυνση. Και αυτό προσπαθώ να κάνω. Προσπάθησα να το κάνω με όλο το κείμενο. Κάποια πολύ σύντομα σχόλια. Δεν είχα την πρόθεση εγώ να πω κάτι αντίθετο προ τα κριτήρια τη Κομπεχάκη. Πολύ καλά λειτουργήσαν, αλλά μετά από 10 χρόνια είμαστε υποχρεωμένοι να ε, δούμε πώ διαμορφώθηκε η όλη διαδικασία. Αυτό προσπαθώ να κάνω. Γι' αυτό περιμένω τις τροπολογίες σας που θα εμπλουτίσουν την έκθεσή μου. Βεβαίως δεν είχα την πρόθεση εγώ να ε, ρίξω αρνητικό φως στα κριτήρια της Κοπεχάης τώρα. συμφωνώ ότι θα πρέπει να ισχύει ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οτιδήποτε μπορεί να βελτιώσει την αξιοπιστή μα είναι καλόδεχτο. Αυτό το οποίο πιστεύω ότι είναι σημαντικό είναι να προσπαθήσουμε στη διαδικασία διεύρυνση να συμμετάσχει όσο περισσότερο μπορεί η κοινωνία των πολιτών. Το έχουμε κάνει, αλλά θα πρέπει ακόμη περισσότερο να το κάνουμε. Και όχι μόνο την κοινωνία των πολιτών των υποψηφίων χωρών μέσω του ΆΙΠΑ 2 διότι μπορούμε σε, να, περι, να δουλέψουμε περισσότερο με την κοινωνία των πολιτών από τις κυβερνήσεις, αλλά και των κρατών μέλων. Θα πρέπει να πείσουμε τους λαούς μας ότι πρόκειται για μία διαδικασία την οποία θα πρέπει να διατηρήσουμε. Ναι, ναι. Τώρα, η όλη διαδικασία σε περίπου εδώ και 10 χρόνια και σε θέματα δικαιοσύνης, όλα τα θέματα που προαναφέρατε σε όλη τη διαδικασία γίνονται όλο και περισσότερο σημαντικά και πρόκειται για ένα τομέα στον οποίο θα πρέπει να επιμείνουμε ευθύ εξ αρχή και όχι στο τέλο, όχι στη μέση τη διαδικασία. Η δυνατότητα απορρόφησης επίσης δεν είναι κάτι το τεχνικό. Δεν είχα την πρόθεση να αποστείλω αυτό το μήνυμα. Είναι όμως ένα γεγονός, μια πραγματικότητα. Κάτι όμως το οποίο έχει και πολύ σημαντική ε, πολιτικές ρίζες αν θέλετε. Πρόσφατα συζητήσαμε στα πλαίσια της Βίρσμα για την ε, πολιτική δυνατότητα παρόφηση των κονδύλων. Και αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Εγώ δεν θέλω να προσθεθούν τα κοινωνικά κριτήρια στα τρία ήδη υπάρχοντα κριτήρια. Δεν υπάρχει εκτιμένο. αλλά υπάρχουν ε, οι γενικοί κοινωνικοί αποδεκτοί με την Ευρωπαϊκή Ένωση κανόνες, στους οποίους θα πρέπει να επιμείνουμε για να συνεχίσουν να ισχύουν. Ευχαριστώ τον κύριο Σεμίνο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που προσπαθούν να βρουν τρόπο συνεννόησης για αυτά τα θέματα, διότι είναι πολύ σημαντικό τα δύο θεσμικά όργανα να προχωρήσουν από κοινού και παραλλήλου για αυτό το θέμα, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Σας ευχαριστώ. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 8 Μαΐου και αναμένω τις συνεισφορές σας. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σε αυτή την πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα συζήτηση. The, uh, chairman... Πριν φύγετε κύριε Μπροκ από την αίθουσα. Μάλλον πριν φύγει. Έκανε μια ενδιαφέρουσα πρόταση, την οποία θα μπορούσαμε να σκεφτούμε, ας πούμε να κάνουμε κάποιες ακροάσεις. Η ακρόαση, ενδιαφέρουσα ιδέα. Και αν γίνει, τότε η προθεσμία που μας βάζετε 8 Μαΐου είναι πολύ σφιχτή για την υποβολή, τελευταία ημερομηνία δηλαδή, για την υποβολή τροπολογιών. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου, κυρία Κοπά, αλλά ίσω θα πρέπει να καθυστερήσουμε. Και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να σκεφτούμε πολύ περισσότερο το θέμα αυτό. Αν υπάρχει λοιπόν δυνατότητα να αλλάξουμε την ημερομηνία, καλό θα ήταν να, την, να, έχουμε μεγαλύτερη προθεσμία δηλαδή. Πρέπει να τελειώσουμε τη συζήτηση. Γιατί περιμένουν στην αδελφή μας για το επόμενο θέμα. Ήθελα να μιλήσω και σε αυτή τη συζήτηση. Ο κύριος ε, Λάνστορφ περιμένει. Περιμένει υπομονητικά. Συμφωνώ με τον Άντριου και χαίρομαι που συμφωνεί και η κυρία Κοπά. Είναι πολύ σημαντική αυτή η έκθεση και πρέπει να τη συζητήσουμε με περισσότερο χρόνο. Επίσης, ε, μπορούμε να διαφωνήσουμε την Κομισιόν. Δεν είναι δεδομένο ότι πρέπει να συμφωνούμε. Και τώρα πάω στην δική μου έκθεση. Το επόμενο σημείο στη μέση διάταξη. Η σύσταση του Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο ε, για την 67η ε, Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Θα τα πω γερμανικά. Βάλτε παρακαλώ τα ακουστικά σας γιατί θα τα πω γερμανικά και θα μιλήσω και αργά για αλλαγή και ορισμένα ε, δευτερεύοντα λέω τώρα μέχρι να βάλετε τα ακουστικά σας. Λοιπόν, φέτος ε, χωρίσαμε τη σύστασή μας σε 7 κεφάλαια. Για ποιο λόγο. Κάθε χρόνο, όπως και πέρσι, είχαμε πάει με αντιπροσωπεία της Επιτροπής Εξωτερικών στη Νέα Υόρκη για να δούμε τις προτεραιότητες και να θέσουμε ακριβώς τα πλαίσια για το τι είναι ρεαλιστικό, εφικτό. Τα 7 κεφάλαια εστιάζουν στο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών. Η παγκόσμια διακυβέρνηση Global Governance παίζει μεγάλο ρόλο και η ειρήνη και η ασφάλεια. Έχουμε ένα κεφάλαιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν στα πλαίσια του ΟΗΕ και τι θέλουμε. Το Κοινοβούλιο εξακολουθεί να πιστεύει ότι η συνάφεια και η προβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να εξασφαλίζεται και ιδιαίτερα η πλήρης εφαρμογή των ψηφισμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας, ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να ε, τηρηθεί και να έχουμε πολύ καλύτερη δυνατότητα συντονισμού στο Συμβουλίο Ασφαλείας. Έχουμε δύο κράτη-μέλη. Γενικά δεν είναι πολύ μεγάλος ο συντονισμός με την Αγγλία και τη Γαλλία και τα μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας λειτουργούν πιο σωστά από τα μόνιμα. Τώρα, η παγκόσμια διακυβέρνηση, στρατηγικό ζήτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε οι εκπρόσωποι ε, των κρατών μελών της Ένωσης αλλά και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συστηματικά να συνεννοούνται και διμερός και πολυμερός εγκαίρως και στη Νέα Υόρκη και του Συμβουλίου Ασφαλείας ευρύτερη μεταρρύθμιση. Δεν έχει να κάνει μόνο με τις έδρες, τον αριθμό και ποιος θα τις κατέχει, τον τρόπο εργασίας και άλλους. Και τα μέτρα ε, της ΑΤΧΟ κομμάδας για την ε, αναζωγόνηση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών είναι σημαντικά αυτά για την παγκόσμια διακυβέρνηση. Ε, κεφάλαιο τρίτο, ασφάλεια και ειρήνη. Ε, ε τώρα, η Peace Building Architecture, αρχιτεκτονική οικοδόμηση της ε, ειρήνης, πρόληψη κρίσεων, διαχείριση κρίσεων πολιτική και στρατιωτική και η αναθεώρηση των πολιτικών δυνατοτήτων. Σημαντικό είναι η συμμετοχή των γυναικών σε όλες ε, τις δράσεις μιας συνευτικής διαδικασίας. Εμπειρικά φάνηκε ότι όπου συμμετέχουν περισσότερο οι γυναίκες ε, βρίσκονται βιώσιμες λύσεις. Επίσης θα πρέπει να συνεχίσουμε ε, περισσότερο στην ανάπτυξη της ευθύνης για προστασία της έννοιας αυτής να ξεκαθαρίσουμε ότι έχει μια πτυχή προληπτική και είναι μια έννοια που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κατά τη διάρκεια της ανοικοδόμησης μετά από μια εμπόλεμη σύραξη. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό και ξέρω ότι εδώ στην Επιτροπή μας μας ενδιαφέρει και ε, κυριάρχησε και όταν δημιουργήθηκε η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης είναι κάποιες μεσολαβητικές δομές, ε, mediation. Η διαμεσολάβηση θα πρέπει να γίνεται καλύτερα με καλύτερες κατευθυντήριες γραμμές, περισσότερους πόρους και καλή συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και το πολιτικό τμήμα ε, του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Τέταρτο κεφάλαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Βεβαίως θα πρέπει να ενισχυθούν οι εθνικές δυνατότητες να τηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Παντού θα πρέπει να παίζει ρόλο αυτό σε όλες τις πολιτικές των Ηνωμένων Εθνών, το mainstreaming, μια παγκόσμια περιοδική αναθεώρηση και στις έκτακτες διαδικασίες θα πρέπει ε, όσο γίνεται νωρίς να κινητοποιείται αυτό. Πέμπτο κεφάλαιο και ιδιαίτερο αφορά την υποστήριξη της δημοκρατίας και πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό με τον καλύτερο τρόπο. Θεωρώ, μαζί με άλλους συναδέλφους, ότι η υποστήριξη για τη δημοκρατία θα πρέπει να υπερβαίνει τις εκλογές και την υποστήριξη παρακολούθηση εκλογών. Και οι κόμματα ε, πολιτικά και κοινοβούλια θα πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο και να τα βοηθούμε προς τα εκεί. Η κοινωνία των πολιτών, είναι ωραία και οι γυναίκες και η πρόθεση των γυναικείων δικαιωμάτων παίζουν ιδιαίτερο ρόλο εδώ. Επίσης, ε, είναι και οικονομική υποστήριξη, αλλά και ε, με στελέχη, ανθρώπινο δυναμικό για την υποστήριξη της δημοκρατίας που είναι βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής και θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται αντίστοιχα σχέση μας με τα Ηνωμένα Έθνη. Το κείμενο για την ανάπτυξη είναι πάρα πολύ στοιχειώδες, θα το διαπίστωσαν συνάδελφοι που το διάβασαν. Ε, σε γενικές γραμμές μας ενδιαφέρει να συνεχίσουμε ε, την καλή συνεργασία με την Επιτροπή Ανάπτυξης. Εκείνοι θα κάνουν γνωμοδότηση και θα συζητήσουμε μαζί τους ποια στοιχεία θέλουν να τονίσουν στην έκθεσή μας. Και ε, τέλος, Λέμε ότι θα πρέπει και το Συμβούλιο να ασχοληθεί με αυτό. Πώς θα δημιουργήσουμε δημόσιο ενδιαφέρον για τα Ηνωμένα Έθνη με συμμετοχή ας πούμε εθνικών κοινοβουλίων. Είναι σημαντικό αυτό ο ΙΕ. Μπορεί να είναι ένας οργανισμός που να χαίρει γενικά κύρους, αλλά αν ρωτήσει λίγο παραπάνω, οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ούτε πώς λειτουργούν τα Ηνωμένα Έθνη, ποιοι πυλώνες υπάρχουν και πώς δουλεύει χρειάζεται μεγαλύτερη κοινοβουλευτική συμμετοχή και αυτό ίσως θα κέρδιζε και μεγαλύτερη υποστήριξη γενικότερα για τα Ηνωμένα Έθνη. Πρακτικές παρατηρήσεις τώρα. Τροπολογίες. Προθεσμία λίγη στις 9 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι, 30 και 31 του μηνό θέλουμε Μαΐου να το συζητήσουμε στην Επιτροπή μας και να ψηφίσουμε. Αρχές Ιουνίου στην αντίστοιχη Επιτροπή του Συμβουλίου θα παρουσιαστεί αυτό. Τέλη Ιουνίου θα αποφασίσει το Συμβούλιο. Χέρι με χέρι λοιπόν και ευχαριστώ και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για τη συνεργασία και για ε, όλη την υποστήριξή σας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και με χαρά θα ακούσω τι έχετε να πείτε και τις παρατηρήσεις σας. Ευχαριστώ. Πρώτος, ο κύριος Πρέντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για δεύτερη φορά είμαι σκιώδης ηγητής του ΑΕΚ για αυτό το θέμα. Και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Λάνστορφ για την ε, ευρεία του έκθεση, για την πλήρη του έκθεση. Θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ΟΗΕ. Για να στέλνουμε μονοσήμαντο μήνυμα, για να είμαστε συνεπείς, για να είμαστε συνεχτικοί, θα πρέπει να συντονιζόμαστε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να έχουμε εσωτερικό συντονισμό. Θα πρέπει επομένω να κατανοούμε μονοσήμαντα την ε, το ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύστημα του ΟΗΕ. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε μεταξύ μα. και μόνο όταν συμφωνήσουμε μεταξύ μα θα καταλάβουν και οι εταίροι, μα μας ότι έχουμε την ίδια άποψη. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μία στρατηγική εφαρμογή του ψηφίσματος. Γιατί υπάρχουν ακόμα διαφορέ στο εσωτερικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σε ό,τι αφορά την ερμηνεία. Και αυτέ οι διαφορετικέ ερμηνείε ακούστηκαν σε διάφορε ε, συνεδριάσεις πιστεύω ότι ήγηκε η ώρα η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να δει πώς εφαρμόζεται το ψήφισμα. Για να δει αν δουλεύει καλά, να μας εξηγήσει τι πρέπει να βελτιωθεί κτλ. Νομίζω ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί το καθεστώς του ειδικού παρατηρητή πριν αναζητήσουμε το καθεστώς του μέλους. Επίσης, τις ευθύνες μας θα πρέπει να τις σκεφτούμε πολύ σοβαρά. Δεν θα πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση για ευθύνες με μια διάθεση προστατευτισμού, γιατί με αυτόν τον τρόπο υποσκάπτουμε την έννοια της ε, ευθύνης για την προστασία, για τη διαμεσολάβηση. Το Συμβούλιο θα πρέπει να έχει μια ευρεία προσέγγιση για την υποστήριξη του εκδημοκρατισμού. Θα ήταν χρήσιμο να αναφέρουμε την υποστήριξη με χρήση των σημερινών χρηματοδοτικών μέσων, ιδίω απέναντι στις, στους ανεξάρτητους ε, ΜΚΟ. Η Αίγυπτος και η Λευκορωσία μας δίδαξαν κάποια πράγματα. Είναι σημαντικές οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις αν θέλουμε να ριζώσει η δημοκρατία. Θα υπάρξουν τροπολογίες του ΕΛΚ για το θέμα αυτό και περιμένω με ανυπομονησία την, μια θαυμάσια συνεργασία με τον εισηγητή μας για την προθεσμία για τις τροπολογίες. Εδώ υπάρχει μια αναφορά στις 26 Απριλίου. Μας δίνετε περισσότερο χρόνο δηλαδή για τις τροπολογίες. Πέστε μας. Γιατί είπατε η 9η Μαΐου είναι η τελική ημερομηνία. Ευχαριστώ. Τελευταίος ομιλητής, η κυρία ο ομιλητη η κυρια Μουνής. Πρόεδρε. Θα μιλήσω ως μέλος Ομάδα εργασία για τα Ηνωμένα Έθνη. Νομίζω ότι η συνάδελφο, η Κορίνα Κρέτσου, που είναι ε, σκιώδης εισηγήτρια τη Ουσιαλιστικής θα συμφωνήσει με αυτό που θα πω και θα ασχοληθεί και είναι περισσότερο με θέματα ανάπτυξη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ακόμη μια φορά και πάλι τον κύριο Λάμστορ για την ε, έκθεση αυτή, την πρόταση αυτή ψηφίσματος που είναι πλήρης και αναφέρεται στην ε, Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και στο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να κάνω κάποιες ε, υποδείξεις και να θέσω τροπολογίε για να το συμπληρώσουμε. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ηνωμένα Έθνη. Νομίζω ότι θα πρέπει να επαναλάβει κάποια σημεία τα οποία υπάρχουν στη δική μου έκθεση, στην οποία λέγεται ότι είχε φιλοδοξίε με τον τρόπο που αποφάνθηκε για αυτά τα θέματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για, την, για τα Ηνωμένα Έθνη. Επίσης, σε θέματα ειρήνη και ασφάλειας γίνεται αναφορά στις γυναίκες, στην ε, περιπτώσεις ε, που υπάρχουν ε, ε, διαφορές και διανόριες. Εκεί αναφέρθηκε ότι υπάρχει η προοπτική της ισότητας των δύο φύλων όταν έχουμε τέτοιου είδους καταστάσεις. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε ότι η συμμετοχή των γυναικών στην επίλυση διαφορών ή η προβληματική των γυναικών θα πρέπει να έχει εγκάρσια ε, διάσταση για τα Ηνωμένα Έθνη. Κυρίως ε, να αναφερθεί και ο ρόλος των γυναικών για τη διασφάλιση της ειρήνης για θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας, ανθρωπιστικής ε, ε, συνδρομής σε θύματα γυναίκες βίας και κακοποίησης και στην τελική φάση που είναι αυτή τη σύναψη των ειρηνευτικών συμφωνιών. Από την άλλη πιστεύω ότι οι σοσιαλιστές μπορούμε να συνεισφέρουμε με πρωτότυπο τρόπο ένα επαναλαμβανόμενο πρόβλημα το ΝΟΗΕ είναι το θέμα της χρηματοδότησης. Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε νέα θεσμικά όργανα, δεν τους δώσουμε τα κατάλληλα κονδύλια για να λειτουργήσουν. Θα ήθελα να προτείνω λοιπόν και θα μιλήσω εδώ για ποσοστά να υπάρχει η δυνατότητα ένα μέρος των συνεισφορών των κρατών μελών να υπάρχει ένα ποσοστό για την ε, ε, χρησιμοποίηση ε, για θέματα που αφορούν τις γυναίκες. Αναφέρουμε στο 0,01% εκαστοτία ποσοστό πολύ μικρό. Τώρα, όσον αφορά την δυνατότητα ε, προστασίας, θα πρέπει να αναφερθούμε σε ένα νέο όρο, ο οποίος χρησιμοποιείται τώρα τελευταία. Responsibility to protect, όπως λέτε. Και θα πρέπει να ζητήσουμε από το Συμβούλιο ως κύριος, ε, ως κύρια προητής ε, τέτοιου θέματα να το συμπεριλάβει και αυτό. Τώρα, για την διαμεσολάβηση. Θα θέλαμε να μιλήσουμε εμείς για προληπτική διπλωματία, να το προσθέσουμε αυτό για να συμπληρωθεί ο τίτλος. Και θα μπορούσαμε και να μελετήσουμε την, τη δυνατότητα να κάνουμε μια κάποια, να δημιουργήσουμε μια κάποια σχέση μεταξύ αυτών το οποίο κάνει για τη διαμεσολάβηση η Ευρωπαϊκή Ένωση και, τα, και ο Και εδώ νομίζω ότι αυτά τα οποία ε, συμπεριλαμβάνονται σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας μπορούν να μας χρησιμοποιήσουν. Επίσης, θα ήθελα να πω το εξής. Τα δυνάμεις του ΟΗΕ να αναλάβουν και την προστασία των ε, διεθνών παρατηρητών κατά τη διάρκεια των εκλογών, της εκλογικής διαδικασίας. Διότι πολλές φορές στο τέλος μιας ειρηνευτικής διαδικασίας που είναι η σύγκληση εκλογών δεν προβλέπει τέτοιου προστασία εκ μέρους του ΟΗΕ και πολλές φορές οι δυνάμεις αυτές οι ειρηνευτικές του ΟΗΕ βρίσκονται χωρίς καμία προστασία. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να το προβλέψουμε. Όσον αφορά το κείμενο τη σύσταση σε σχέση με την κατάσταση στην Μέση Ανατολή θα πρέπει να ανακτήσουμε την ε, πρωτοβουλία του 74 του ΟΗΕ να έχουμε μία μέση Ανατολή χωρίς πυρηνικά όπλα. Δεδομένου ότι υπάρξει πολλαπλασιασμός των πυρηνικών όπλων, είναι ανισχυτική η κατάσταση που διαγράφεται σήμερα στο Ιράν. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να επαναλάβουμε εμείς αυτή την πρωτοβουλία της, ε, του ΟΗΕ για να έχουμε μία μέση Ανατολή χωρίς πυρηνικά όπλα. Και τελικά... Νομίζω ότι ίσως αυτό ήταν ε, ε, κάτι το που το παρέλειψαν να αποσταλεί η σύσταση αυτή και στην ε, το εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική. Ευχαριστώ. Είμαστε στην αρχή της διαδικασίας. Βεβαίως χαίρομαι για τη συνεργασία που έχει αποδειχτεί χρήσιμη. Ενδιαφέρουσα υποσώστοση για την εργασία των γυναικών στα Ηνωμένα Έθνη. Το είπε και η κυρία Μουνίθ ότι ε, έχει πρόβλημα στελέχωσης η υπηρεσία γυναικών, UN Women. Να το συζητήσουμε αυτό μεταξύ των εισηγητών, αν θέλουμε να το συζητήσουμε, και των σκιωδών. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες παρεξηγήσεις για την προθεσμία. Δεν είναι 26 Τετάρτου, αλλά η 9η Μαΐου. 9η Μαΐου για τις τροπολογίες και μετά θα μπούμε στη διαδικασία της συζήτησης για να ε, το φέρουμε σε αίσιο πέρας. Δυστυχώς πρέπει να φύγω. Αργήσαμε να συζητήσουμε το θέμα μου, αλλά θα το ξανασυζητήσουμε, δεν είναι τελευταία φορά. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Προθεσμία λοιπόν κατάθεση απολογιών 9η Μαΐου. Να σας κάνω και μια πρόταση να το συζητήσουμε και με την κυρία Κοπά. Αποφασίσαμε για τις 8 Μαΐου. Αλλά μετά τη συζήτηση ε, που κάναμε, όταν έρθουν τροπολογίες, θα πρέπει η κυρία Κοπά ενδεχομένω να κάνει και ένα δεύτερο σχέδιο έκθεσης μετά από τις τροπολογίες για να το συζητήσουμε μετά την ακρόαση που θα κάνουμε κτλ. Για να μην πάμε τον Ιούνιο στην Ολομέλεια, αλλά τον Ιούλιο. Συμφωνείτε? να αφήσουμε την 8η Μαΐου, αλλά με τη δυνατότητα μετά την ακρόαση να ξαναγράψει την έκθεσή της η κυρία Κοπά. Αλλά δεν θέλω να το αποφασίσουμε χωρίς να το έχω συζητήσει προηγουμένως μαζί της. Αλλά ε, από την πορεία της συζήτησης αυτό προέκυψε. Δεν διαφωνεί κανείς από ό,τι βλέπω. Ευχαριστώ πολύ. Και πάμε στο επόμενο θέμα της μέσης διάταξης και τελευταίο μάλλον.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 I would like to introduce you, Λοιπόν, θα ήθελα να σας συστήσω τον κύριο Γιάννη Κάρτινς, ε, αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή για την Επικοινωνία και την Ενημέρωση της UNESCO. Θα μας μιλήσει σχετικά με τις δραστηριότητες της UNESCO στη Νότιο Μεσόγειο. Σημαντικότατο ζήτημα, διότι συνεργαζόμαστε ε, εκεί και μάλλον και λεφτά θα στέλνουμε από την Ένωση. Έτσι δεν είναι. Πάντως η συνεργασία μας με τους οργανισμούς του ΟΗΕ είναι εξαιρετική σημασία. Και θα ήθελα να παρακαλώ τον κύριο Κάρκλινς να λάβει το λόγο. Παρακαλώ και σα ευχαριστώ που ήρθατε. Thank you, Mr. And, Ευχαριστώ, uh, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία μέρους της UNESCO να παρουσιάσω σύντομα τις δραστηριότητε μας στον τομέα της έκφρασης της ελευθερίας, της ανάπτυξης των ΙΕ στη Βόρεια Αφρική και τα Αραβικά κράτη και την Νότιο Μεσόγειο. Η UNESCO είναι πιο γνωστή στο... για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Όμως εδώ και πολλά χρόνια η UNESCO ασχολείται πολύ ενεργά με θέματα ελευθεροτυπίας έκφρασης και ελευθερίας έκφρασης, και ελευθεροτυπίας. Και ε, προωθούμε διάφορες δράσεις καταρχάς μια συστημική προσέγγιση σε θέματα ελευθεροτυπίας μέσω νομοθεσίας. Εκεί συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη για να τα βοηθήσουμε να προσαρμόσουν τα ΜΜΕ ε, και τους νόμους για την ελευθεροτυπία, να υπάρξει πρόσβαση σε πληροφόρηση και να σεβαστούν τα διεθνή πρότυπα σχετικά. Αυτές ήταν οι πρώτες δράσεις της ε, UNESCO μετά την Αραβική Άνοιξη στην Τινησία, στην Αίγυπτο και στην Ιορδανία όμως. Και τώρα ετοιμαζόμαστε να δράσουμε με αντίστοιχες δράσεις με τις νέες ε, λιβικές αρχές. Η μεγάλη προβολή της δουλειάς της UNESCO ε, είναι η, μέρα, η Παγκόσμια Μέρα ελευθεροτυπίας, ε, κάθε χρόνο στις 3 Μαΐου. Πριν από 21 χρόνια, 3 Μαΐου, ε, κάποιοι Αφρικανοί δημοσιογράφοι έκαναν μια δήλωση και ζήτησαν να υπάρξει μια τέτοια μέρα παγκόσμιας ελευθεροτυπίας. Παγκόσμια μέρα ελευθεροτυπίας. Αυτή την μέρα τη συνδέουμε με την απονομή ενός βραβείου σε εφημερίδα ή δημοσιογράφο, ο οποίος έχει συνεισφέρει σε... στην αποκατάσταση ελευθεροτυπίας οπουδήποτε στον κόσμο. Στο φέτος δώσαμε το βραβείο αυτό στον Ανούλα Φατουλάιεφ ε, από το Αζερμπαϊτζάν. Και στην Καρθαγέννη Καρχιδόνα, συγγνώμη, θα γίνει η γιορτή αυτή στη Δινησία, όπου θα είναι παρούσες και οι αρχές και ο Πρωθυπουργό. Ε, συνήθως αυτοί οι εορτασμοί συνοδεύονται από μία διάσκεψη. Ε, κάθε χρόνο η διάσκεψη αυτή συζητάει ένα συγκεκριμένο θέμα, διαφορετικό. Φέτος θα συζητήσουμε τις νέες φωνές στην ελευθεροτυπία ε, του τύπου που βοηθούν για το μετασχηματισμό των κοινωνιών μας θα αναλύσουμε το ρόλο των ΜΜΕ στις ε, κοινωνίες ε, σε μετασχηματισμό, το ρόλο της νεολαίας και τις νέες τεχνολογίες ε, στον κοινωνικό μετασχηματισμό. αλλά σημαντικό είναι να μιλήσουμε και για το ρόλο των βουλευτών για να εξασφαλίσουν την ελευθερία της έκφρασης, την ελευθεροτυπία στις χώρες που βρίσκονται σε μεταβατική φάση. Οι δραστηριότητε της UNESCO στην περιοχή Μένα ε, έχω σε σκοπό να δημιουργηθεί το δυναμικό δημιουργία ε, σχολών για τους δημοσιογράφους, την κατάρτιση δημοσιογράφων ε, και η πρώτη δράση που προωθήσαμε μετά την αναταραχή ήταν να εκπαιδεύσουμε δημοσιογράφους στην Αραβική Άνοιξη για την, να μας μιλήσουν για τις εκλογές. Γιατί ήταν σημαντικό ότι μετά από δεκαετίες με καθεστώτα όπου μία ήταν η αλήθεια, μία ήταν η φωνή, θα έπρεπε να εκπαιδεύσουμε νέους δημοσιογράφους για τον πλουραλισμό και να τους πούμε ότι υπάρχει, ότι μπορεί να έχουν διαφορετικές απόψεις όσοι κατεβαίνουν σε εκλογές. Το μέσο που χρησιμοποιεί η UNESCO ε, στις χώρες όπως η Αίγυπτος ή η η Ισία είναι ε, μια μεθοδολογία που θα βασίζεται σε δείκτες. ξεκινήσαμε τέσσερα χρόνια πριν, έχουμε, την έχουμε εφαρμόσει τη μεθοδολογία σε διάφορες χώρες και μας επιτρέπει αυτή η μεθοδολογία να αναλύσουμε και να εντοπίσουμε τα κενά τα οποία θα πρέπει να καλυφθούν στον τομέα της και προωθούμε κάποια project στην Τινησία, στην Αίγυπτο και στην Ιορδανία. Στην περιοχή Μένα δηλαδή. Η συνεργασία με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ σημαντική για την UNESCO. Και αμέσως μετά τα γεγονότα ήρθαν σε επαφή διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μα είπαν ότι θέλουν να χρηματοδοτήσουν διάφορα project. Το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Σουηδία. Αυτές ήταν οι τρει πιο δραστήριε και πιο γενναιόδορες ε, χώρες, οι πιο γενναιόδοροι δωρητέ. και προωθούν κάθε μία διαφορετικά project. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή εξετάζει κάποια πιο μεγάλα project για όλη την ε, περιοχή την δημιουργία ενός κρατικού ραδιοσταθμού και αν τα πράγματα εξελιχθούν όπως περιμένουμε, η UNESCO θα είναι η βασική υπηρεσία εφαρμογής, μέσω της οποίας θα, θα εφαρμοστεί αυτό το project. Η μεγάλη σημασία που δίνει η UNESCO στην ασφάλεια των ε, δημοσιογράφων και στην καταπολέμηση της ατιμορρησίας είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί δεν μπορούμε να χτίσουμε μια ζωντανή κοινωνία, να απειλούμε τους δημοσιογράφους αν τους ε, παρενοχλούμε ή τους σκοτώνουμε. Το Σεπτέμβριο του 2011 οργανώσαμε μια ε, συνάντηση της, του ΟΗΕ για την ασφάλεια των δημοσιογράφων που οδήγησε σε ένα σχέδιο δράσης για την ασφάλεια των δημοσιογράφων και η UNESCO είναι η βασική υπηρεσία του ΟΗΕ που ασχολείται με αυτό το θέμα της ασφάλειας των δημοσιογράφων και την καταπολέμηση της ατιμορρησίας. Υπάρχουν διάφορα σημαντικά στοιχεία σε αυτό το σχέδιο δράσης με σκοπό μια καλύτερη συνεργασία των διαφόρων υπηρεσιών του ΟΗΕ για αυτά τα θέματα ε, και απευθύνεται στα κράτη-μέλη. Ένα ζήτημα είναι. Το Συμβούλιο Ασφαλείας μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο σε θέματα ασφάλειας των δημοσιογράφων, πέρα από τις ε, περιοχές όπου υπάρχει πόλεμος και σειράξεις. Το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας 1738 είναι ε, το βασικό μας κείμενο για τέτοια θέματα ασφάλειας δημοσιογράφων σε περιοχές πολέμου. Αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι οι περισσότεροι δημοσιογράφοι σκοτώνονται όχι σε θέατρα πολέμου, αλλά εκτός. Και αυτό είναι βασικό θέμα του σχεδίου δράσης μας. Φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση καλό θα ήταν να εμπλακεί στο θέμα αυτό και οι ευρωβουλευτές να συμμετάσχουν στη συζήτηση γιατί καθήκον της κοινωνίας είναι να προκαλ... να προστατεύσει τους ε, δημοσιογράφους και των κυβερνήσεων καθήκων, αλλά βεβαίως και της κοινωνίας. Γιατί θα πρέπει να υπάρχει ε, μια, ένα πνεύμα έτσι ανοχής, ένα πνεύμα έλλειψη μυσαλλοδοξίας απέναντι στους δημοσιογράφους. Τώρα για την ημέρα, ε, Παγκόσμια ημέρα ελευθεροτυπίας που φέτος θα γιορταστεί στην Τινησία όπως σας είπα. Καλό και τους ευρωβουλευτές στην Τίνιδα στις 3 Μαΐου για να γιορτάσουμε την Παγκόσμια ημέρα ελευθεροτυπίας για να συζητήσουμε θέματα του ρόλου των ΜΜΕ στις ε, κοινωνίες που βρίσκονται σε μετάβαση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με χαρά θα απαντήσω οποιαδήποτε ερώτηση έχουν οι ευρωβουλευτές. Ah, Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Γκάλερ στα λετωνικά, στη μία φράση που ξέρω. Ε, σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας και γενικότερα πρώτα πρέπει να σας πω ότι με θετικά που η UNESCO δραστηριοποιείται τόσο πολύ σε αυτό το τόσο ειδικό θέμα. Διότι βεβαίως η UNESCO έχει και κάποια κράτη-μέλη που δεν διακρίνονται, δεν είναι πρωταθλητές στην ελευθεροτυπία. Και χαίρομαι που εσείς δραστηριοποιήσετε τόσο πολύ και με τρόπο τόσο ε, συγκεκριμένο. Γιατί υπάρχουν κράτη-μέλη στην UNESCO που δεν είναι πρωταθλητές της ελευθεροτυπίας. Και αυτή η διαδικασία τώρα στη Βόρεια Αφρική μπορεί ε, να μην είναι δυνατή αλλού. Ίσως στη Ρωσία ακόμα, αλλά στην Κίνα σίγουρα όχι. Λοιπόν, σας εύχομαι ε, καλή τύχη εκεί που σας επιτρέπουν να δραστηριοποιήσετε. Ενδιαφέρομαι πάρα πολύ για την περιοχή γιατί ήμουν επικεφαλής ε, της αποστολής παρατήρησης των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Τινησία και βεβαίως ε, ασχοληθήκαμε και με το θέμα της ελευθερίας του τύπου και τον τρόπο με τον οποίο παρουσίασε ο τύπος τις εκλογές. Σε αυτή την όλη ιδιαίτερη κατάσταση ε, βεβαίως σε πολιτικό επίπεδο ήταν από το παλιό καθεστώς. Παρ' όλα αυτά υπήρχε μια ειδική κατάσταση και δεν ξέρω αν μπορεί να αντιμετωπιστεί σωστά. Είχαμε δημοσιογράφους που ήταν πρώην πιστή του καθεστώτος και παρέμεναν στα κρατικά μέσα ενημέρωση και σε κάποιες εφημερίδες και άλλους δημοσιογράφους που ήταν στην αντιπολίτευση πριν. Και ποιο πρόβλημα είδαμε εμείς ανεξάρτητα από ποια τοποθέτηση είχε ο καθένα της παλιάς φρουρά ή της νέα και πέρα από το γεγονός που αναφέρατε κατά πολέμηση της ατιμορρησία και προστασία των δημοσιογράφων. Εκεί που θα μπορούσατε ενεργά να συμμετέχετε είναι να κάνετε σεμινάρια, μαθήματα, διασκέψεις, ξέρω εγώ για να αυξηθεί και αναβαθμιστεί ε, η επαγγελματική δεοντολογία της δημοσιογραφίας. Αυτό συμβαίνει σε πολλές χώρες σε μετάβαση. Δεν υπήρχε ελευθερία πριν, οπότε προσπαθούσε ο καθένας ή ορισμένοι να δείξουν ένα οπορτουνισμό, ε, να κεροσκοπήσουν ή απλώς ήταν στην παρανομία τα έντυπα, αλλά τώρα είναι όλα ελεύθερα και ο κόσμος πιστεύει ότι ε, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, να επικρατεί ασυνδοσία, ο διάφορες φήμες που ακούν ε, τις δημοσιεύουν ως γεγονότα χωρίς να τα διασταυρώνουν ε, στις εφημερίδες, να μην γίνουν σχόλια και ειδήσει ε, και στο ηλεκτρονικό τύπο, στα οπτικοακουστικά μέσα. Και σας ερωτώ και σας παρακαλώ, δεν ξέρω, μπορεί και να το κάνετε ήδη, να ε, επικεντρωθείτε εκεί. Ελευθεροτυπία ναι, αλλά με κάποια δεοντολογία να είναι πιο επαγγελματίε οι δημοσιογράφοι και όχι αυτή η ασυδοσία που επικρατεί. Έτσι ώστε να ξέρουν ότι κάνουν τη δουλειά του για του πολίτε του ίδιου. και να μπορούν οι πολίτε να εμπιστεύονται τα νέα μέσα. Γιατί τι νόημα έχει να αποστοσιοποιηθεί κανεί από ε, ε, τα παλιά μέσα του καθεστώτος και να χαίρει τις ελευθερίες και ξαφνικά να ανακαλύπτει ότι και τώρα με τους νέους καιρούς ό,τι γράφεται δεν είναι απαραίτητο αλήθεια. Τι κάνετε εσεί γι' αυτό. Ε, κυρία Γκόμες, ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίαση, για την παρουσίαση που κάνατε για κάποιον που έχει εμπειρία δικτατορίας, κατανοώ πόσο βασικό και θεμελιώδες είναι να έχουμε την ελευθερία έκφρασης και την ελευθεροτυπία για να εξασφαλίσουμε τη δημοκρατία. Και θα έλεγα ότι πρόκειται για την πρώτη από τις ελευθερίες. Και ο, ο ρόλος των μέσων ενημέρωση είναι πρωταρχής σημασίας. Πριν να γίνουμε μέλη της Ευρωπαϊκή στη χώρα μου πιστεύαμε ότι κάποια στιγμή θα γυρίζαμε πίσω εάν δεν μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε την ελευθερία του τύπου. Και αυτό είναι κάτι το φυσικό. Χαιρετίζω λοιπόν τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η UNESCO και το ότι ευαισθητοποιεί για την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όποια και είναι η κουλτούρα του καθενός. Όντως είναι οικουμενικά, οικουμενικό θέμα και επίτευξη η ε, σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τούτου λεχθέντος θα ήθελα να σας ζητήσω το εξής. Μπορείτε να μας πείτε λεπτομερέστερα τι ακριβώς κάνετε στη Λιβύη, δεδομένου ότι απαιτείται εκεί μεγάλη δουλειά να γίνει και αυτό είναι και ένα από τα νέα θέματα που σας έχουν ανατεθεί στα πλαίσια της ε, διάσκεψης του Παρισιού. Πώς μπορείτε να έρχεστε σε επαφή με την Αφρική γενικότερα, πέραν των ορίων της περιοχής μένα, διότι βλέπουμε να υπάρχουν τρομερά προβλήματα και δεν βλέπουμε να κάνει το σωστό η Πώς μπορείτε να εξηγήσετε ε, το βραβείο Μπιάνγκ που αποφασίστηκε από την UNESCO. Ο Μπιάνγκ είναι ένας από τους πιο σκληρούς δικτάτορες και το ότι έχει χρήματα δεν σημαίνει ότι μπορεί να εξαγοράσει την UNESCO για να του απονείμει ένα βραβείο. Πώς ασχολείται με τέτοιου θέματα λοιπόν η UNESCO. Επίσης θα ήθελα να σας ερωτήσω πώς ε, συνεργάζεστε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι η Αιθιοπία είναι η, από τις χώρες όπου υπάρχει η πιο απάνθρωπη και σκληρή παραβίαση των δικαιωμάτων δημοσιογράφων. Εκεί κρατούνται, είναι φυλακισμένοι χιλιάδε δημοσιογράφοι και υπάρχουν εκατοντάδε και άντρε και γυναίκες που όντω είναι στην φυλακή για γελίου λόγους και κατηγορίες που δεν έχουν καμία σχέση με τις υποχρεώσεις τη χώρα αυτή. Τελικά για το Αζερβαϊτζάν. Χαιρετίζω το ότι απονέμεται βραβείο στους ε, δημοσιογράφους ε, του Αζερμπαϊτζάν. Διότι προβλέπεται και η Eurovision να λάβει χώρα εκεί. Και ελπίζω ότι όντως θα γίνουν σαν τα πράγματα και δεν θα διώκεται εφ' κανείς. Νομίζω ότι είναι μεγάλο γεγονός το ότι γίνεται εκεί η Eurovision και αυτό που κάνετε είναι σημαντικό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Καρτίνς, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους Ευρωβουλευτές για τις ερωτήσεις που μας έκαναν. Κύριε Γκάλερ, Συμφωνώ απολύτως μαζί σας ότι ο επαγγελματισμός των δημοσιογράφων είναι πρωτοϊκής σημασία για τις χώρες αυτές που βρίσκονται σε μεταστηματικό στάδιο. Πρώτα απ' όλα προσπαθούμε να, προσπαθήσαμε να δούμε ποιες ήταν οι επιτακτικές ανάγκες των δημοσιογράφων ε, μετά την, ε, τα γεγονότα πριν να οργανωθούν εκλογές και αναφέρομαι στο πολιτικό επίπεδο και στην ε, Αίγυπτο και στην Τινησία. Δημιουργούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να συνεργαστούμε με τα διάφορα θεσμικά όργανα ότι εμείς δεν έχουμε την αρμοδιότητα αν θέλετε να ασχοληθούμε απευθείας με θέματα κατάρτισης. Προσπαθούμε λοιπόν να δημιουργήσουμε τους θεσμούς που θα αναλάβουν αυτό το έργο. Και νομίζω ότι στο θέμα αυτό μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Πριν από τέσσερα χρόνια η UNESCO έκανε ένα πρωτότυπο πρόγραμμα για την κατάρτιση των δημοσιογράφων και λάβουμε υπόψη ότι μπορεί να γίνει σε επίπεδο σχολείων επί τόπου. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο στην περιοχή ενέκριναν 60 σχολεία σε 50 χώρε, σε 15 χώρες με συγχωρείτε, στο Μαρόκο και στην Αίγυπτο. Ένα από τα θέματα με τα οποία επίσης θα ασχοληθούμε την ημέρα του εορτασμού της ελευθεροτυπίας είναι το θέμα της ηθικής και του επαγγελματι... της επαγγελματικής ε, δημοσιογραφίας, διότι είναι σημαντικά. Ακόμη δεν εργαζόμαστε στην Λιβύη. Το λέγω αυτό για να απαντήσω στο ερώτημα της κυρίας Γκόμες, διότι η κατάσταση ε, σε σχέση με την ασφάλεια δεν είναι ακόμη ότι καλύτερο, αλλά θα το κάνουμε όσο νούπο. Θα δούμε με την Αίγυπτο, την Ιορδανία και την Τινησία τι ακριβώς γίνεται, ποιοι είναι οι δείκτες που θα μας ε, ε, οδηγήσουν σε δράση και εκεί. Προς το παρόν όμως πρέπει να πω ότι δεν έχουμε τους πόρους για να αρχίσουμε μια κάποια δραστηριότητα στην Λιβύη, διότι ακόμη κανένας δωρητής δεν έχει εκφράσει ενδιαφέρον για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων, αλλά αναμφίβολα Κάποιος θα ενδιαφερθεί, ίσως ο παραδοσιακό γείτονας Ιταλία. Τώρα, μία από τι δραστηριότητε μας είναι η ελευθερία της έκφρασης και εκεί έχουμε για την ανάπτυξη των μέσων ε, συνεργασία μέσω διευρυντικών προγραμμάτων και στα πλαίσια αυτών των προγραμμάτων το 50% των δραστηριοτήτων αφορούν διάφορα projects στην Αφρική. Και περισσότερο από 100 εκατομμύρια δολάρια έχουν δοθεί σε περίπου 1500 σχέδια, μισά από τα οποία, να μην πω περισσότερα, η πλειοψηφία προβλέπεται για την Αφρική. Επίσης με την ε, Αφρικανική Ένωση είμαστε σε επαφή και έχουμε για την ελεύθερη ελευθερία της έκφρασης ένα πρόγραμμα συνεργασίας. Συνεργαζόμαστε για την προώθηση της ελευθεροτυπίας με κάποιες κυβερνήσεις της Αφρικής, κυρίως για την πρόθεση της σχετικής νομοθεσίας, την πρόσβαση στην ενημέρωση. Με αυτό ασχολούμαι σε αυτό το τομέα στην Αφρική σήμερα και όσον αφορά την ανάπτυξη των μέσων ενημέρωση, την κατάρτιση των δημοσιογράφων, Έχουμε και διάφορα κέντρα αριστεία σε διάφορα σχολεία στην Αφρική. Έχουμε περίπου 20 σχολεία τέτοια και κέντρα ε, αριστεία, κέντρα αριστείας και οι δραστηριότητες βασίζονται σε πρωτότυπα προγράμματα τα οποία έχουμε αναπτύξει στην UNESCO για την κατάρτιση Αφρικανών δημοσιογράφων. Τώρα, όσον αφορά το βραβείο Μπιάνγκα, αυτό δεν έχει καμία σχέση με την ε, ελευθερία της έκφρασης. Αυτό είναι κάτι το οποίο προτάθηκε από την αντιπροσωπεία της Γουινέσης σημερινού, εγκρίθηκε από όλα τα κράτη-μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου με συνένεση το 2009 και από τότε το Διοικητικό Συμβούλιο ασχολείται με το θέμα αυτό. Ασχολήθηκε μάλιστα πολλές φορές και πρέπει να σας πω ότι είχαμε πάρα πολύ έντονες συζητήσεις μεταξύ των διαφόρων αντιπροσωπιών. Δεν βρήκαμε συνένεση και στην τελευταία συνεδρίαση ψηφίσαμε για το θέμα αυτό. Άλλαξε το όνομα του βραβείου αλλά παρόλα αυτά δεν μπορέσαμε να καταλήξουμε και σε ομοφωνία. Και με πλειοψηφία είπαμε άλλαξε το όνομα του βραβείου. Τώρα να αφορά το Αζερμπαϊτζάν και άλλες χώρες. Η UNESCO ο, Γενικός Διευθυντής καταδικάζει δημοσίως το γεγονός ότι συστηματικά και οργανωμένα δολοφονούνται δημοσιογράφοι. Όσον αφορά τα άλλα θέματα που αφορούν την ελευθερία του τύπου και των δημοσιογράφων. Δεν κάνουμε πάντα δημόσιες παρεμβάσεις ή δηλώσεις. Κάνουμε πιο στοχευμένες δράσεις Είμαστε σε συνεργασία με κυβερνήσεις, με επαγγελματικές οργανώσεις που πιστεύουν ότι η συνεισφορά της UNESCO θα μπορούσε να βοηθήσει την κατάσταση και να προωθήσει την ελευθερία του τύπου. Και αυτό βεβαίω έχει σχέση με τις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες, όπου έχουμε αναλάβει δράση για την ελευθερία του τύπου. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε. Κι εγώ. Δεν ήξερα όλα αυτά τα πρακτικά που κάνει η UNESCO σε αυτούς τους τομείς. Αρκεί και μόνο γι' αυτό το λόγο να προσπαθήσουμε να συνεργαζόμαστε περισσότερο για αυτά τα θέματα. Γιατί ε, προσπαθούμε να ομοθετήσουμε και εμείς για θέματα τύπου και μας ενδιαφέρουν και αυτά που κάνετε και στην Τινησία και στην Αίγυπτο και το, σε δημόσιες ραδιοτηλεοράσεις. Προσβλέπω σε μια συνεργασία μαζί σας και όπου μπορεί να βοηθήσει το κοινοβούλιο, τα κοινοτικά προγράμματα για να ενισχύσουμε και τις εξουσίες και αρμοδιότητες που έχουμε ως κοινοβούλιο σε αυτό το θέμα. Νομίζω λοιπόν θα ήταν καλό να προχωρήσουμε έτσι σε αυτό το δρόμο της συνεργασίας. Μου λέγουν ότι το 2013 θα γιορτάσετε την Παγκόσμια ημέρα ελευθεροτυπίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Α, διερευνάτε αυτή τη δυνατότητα. Να σας βοηθήσουμε να το πετύχετε τότε. Για το 2013 έχουμε και την επέτειο των 25 ετών του βραβείου Ζαχάροφ. Στην αρχή ήταν για την ελευθερία του λόγου πριν για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα μπορούσαμε να τα συνδυάσουμε αυτά τα δύο. Νομίζω είναι μια θαυμάσια ευκαιρία για να το διερευνήσετε και αυτό πώς μπορούμε να το συνδυάσουμε και να αξιοποιήσουμε και τις δύο επαιτίους ε, για να το επιτύχουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και με χαρά σας ξαναδούμε σύντομα και να συνεργαστούμε γόνιμα. Ευχαριστώ. The meeting συνεδρίασης.